Colleagues, the... Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε και πάλι και ας περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι το θέμα αριθμός 17 με 19 που είναι το πακέτο για την κυκλοφορία οχημάτων 17, 18 και 19. Στις 13 Μαΐου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Το λέω ήδη από τώρα, να το ξέρετε, να το ξεχάσω μετά. Θα αρχίσω με τον κύριο Κουν για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων ε, οχημάτων και των ρημουλκούμενών τους. Θα ξεκινήσω με τους τρεις συγητές, μετά δηλαδή η κυρία Σενολοβά και η κυρία Σαβισάρ. Και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους. Ο κύριος Κούν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών δεν έχει υπεράσει. Έχουμε 300 τροπολογίες για το περιοδικό τεχνικό έλεγχο. 29 για τα τεχνικά παραρτήματα, υπόλοιπε για τα άρθρα. Κάποια κεφάλαια προσπαθώ να τα επεξεργαστώ ώστε να δώσω έμφαση περισσότερο στα θέματα στα οποία μπορούμε να επιδιώξουμε συμβασμούς. Νομική ε, πρόταση, νομοθετικό κείμενο, ε, φύση, δηλαδή κανονισμός ή οδηγία, όπου κάποιοι συνάδελφοι όπως ο κύριος Κουμουξάκος, ο κύριος Χίκινς, Βαντάλεν και λοιποί, Σάντσες, Σμιτ, ζητούν να προτιμηθεί ο, ε, αντί για τον κανονισμό η οδηγία, τον κανονισμό έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πάντως το σημαντικό είναι να προσδιοριστούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και να περιγραφούν. Επίσης, στο άρθρο 2.1 υπάρχει μια πρόταση, μια προσπάθεια να βρεθεί ε, συνενετική συμβαστική λύση. Μία πρόταση για διαγραφή τη σχετική για τα οχήματα μέχρι 750 κιλά, θα κοιτάξω ε, να επαληθεύσει αν μπορούμε να την ε, εισαγάγουμε και μέχρι τους 3,5 τόνους που είναι ένα ζήτημα βέβαια γενικό οδικής ασφάλειας και αρκετά περίπλοκο, θα πρέπει να το κοιτάξουμε προσεκτικά. Οι τροπολογίες σχετικές ε, με τον αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογής των σκούτερ, δίκυκλων δηλαδή, μοτοποδηλάτων, υπάρχουν. Υπάρχουν προτάσεις από τους συναδέλφους από την Ολλανδία, από τη Γαλλία. όπου νομίζω ότι θα πρέπει να συνοηθούμε μέχρι ε, πού θα χαράξουμε ακριβώς τη γραμμή σε σχέση με τα μικρότερα ε, μηχανοκίνητα, δίκυκλα, οχήματα. Που, ποια θα βγαίνουν από το πεδίο εφαρμογή και ποια όχι. Θα πρέπει να δούμε τα ε, πιο βαρέα από αυτά τα οχήματα ε, που μπορεί να αποτελέσουν ε, κίνδυνο για την οδική ασφάλεια και αναλόγως να βρούμε μια συμβαστική λύση για το, τα τρακτέρ, τα γεωργικά μηχανήματα πάνω από 40 χιλιόμετρα την ώρα μπορούμε να βρούμε μια λύση μπορούμε να ορίσουμε δηλαδή ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογής στο, χώρο, στο χωράφι, στο εργοτάξιο κτλ. μέσα δεν θα υπάγονται, δεν υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο, αλλά όταν θα βγαίνουν στους δρόμους, ε, όταν θα μεταφέρουν βαρέα φορτία, θα μπορούν να επαχθούν στον, τεχνικό, στον έλεγχο ε, των συνθήκων. Μετά έχουμε τις τροπολογίες 116-118 που θα συζητήσουμε με τους σκιώδεις και θα διαπραγματευτούμε στο θέμα αυτό για τους ελκυστήρες. Στα ιστορικά οχήματα, αντίκες, Έχουμε 20 τροπολογίες. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις. Έχουν καταθέσει από όλες ομάδες, συνάδελφοι, τις τροπολογίες αυτές για να προσδιοριστούν επακριβώς τα κριτήρια και να υπαχθεί η τελική κρίση στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. τελική κρίση για το τι σημαίνει ιστορικό, ιστορική αξία και σημασία όχημα, δηλαδή αν θα μετράει μόνο η ηλικία του ή και η τεχνική του εικόνα, κατάσταση, η εμφάνισή του, όλα αυτά. Εάν θα μπουν και άλλοι ορισμοί. Για, τον, για το άρθρο 3 στους ορισμούς, τι σημαίνει roadworthiness test, δηλαδή ε, έλεγχος ε, ε, δυνατότητας να κυκλοφορεί στους δρόμους, τεχνικός έλεγχος, τι θα οριστεί, πώς θα περιγραφεί αυτό. Θα βρούμε πιστεύω μια λύση σύμφωνη με τις προτάσεις, ώστε να είναι σαφής. Πρόσβαση στο άρθρο 4, πρόσβαση στα δεδομένα του ε, παραγωγού. Νομίζω ότι εδώ οι περισσότεροι συνάδελφοι ε, μας υποστηρίζουν ε, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα, να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα και, την, και η επιθεώρηση, ώστε ο επιθεωρητής να μπορεί να έχει τα στοιχεία όλα στη θέση του. Η επιλογή. Λέω ότι θα πρέπει να έχουμε μία περιοδικότητα 4-2-2 ως προς τα χρόνια. Οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν υποστηρίξει την ιδέα αυτή, τις διετίες δηλαδή για, την, ε, για, τον, για τον έλεγχο. Επιλογή για τα για τα προσωπικής χρήσεως και τα μικρά βαν της πρώτης κατηγορίας αυτά που έχουν περισσότερα διανυθέντα χιλιόμετρα θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάγονται σε πιο τακτικούς ελέγχους, άρα εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Και πάλι στα χιλιομετρικά, στο κριτήριο της χιλιομετρικής απόστασης που επιλέγεται η Επιτροπή το έχει προτείνει μετά την πρώτη αδειοδότηση 4 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα ως διανηθής απόσταση ε, ε, μετά την οποία πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά ο πρώτος τεχνικός έλεγχος. Γκρός, Τυρόν, Τίτσαο, Κοχ, εγώ το είχα αφήσει το, το θέμα αυτό της χιλιομετρικής απόστασης από την έκθεσή μου, το επαναφέρουν όμως οι συνάδελφοι και εισάγουν πάλι την ιδέα ενός ε, πρώτου τεχνικού έλεγχου μετά από, την, ε, ε, μετά από συγκεκριμένο αριθμό χιλιόμετρων. Πάντως θα το δούμε, αλλά ένα χιλιομετρικό κριτήριο φέρει τον κίνδυνο της, του πειράγματος, όπως θα λέγαμε, της επέμβασης των ταχογράφων. Και μετά στον τομέα του άρθρου 12 και τον διαχωρισμό μεταξύ της ε, αποκατάστασης ή της διόρθωσης και της ε, επιθεώρησης. Ε, έχουμε μια τροπολογία 75 και άλλες. Ο κύριος Σκόφε, παραδείγματι, μεταξύ άλλων, λένε ότι θα πρέπει η διόρθωση να γίνεται με βάση τους, τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά να διεξάγεται από άλλον, από άλλο συνεργείο. Οι συνάδελφοι Πίρκερ, Φώστερ, Φαντάνιελ, Μπράιν Σίμψον. Φαντάζομαι στηριζόμενοι και στην εμπειρία των δικών τους ε, των οικείων κρατών μελών, λένε ότι μπορεί να γίνεται η πιστοποίηση στο εργαστήριο το οποίο θεωρείται επαρκώς ε, ανεξάρτητο ώστε να προσφέρει το σχετικό πιστοποιητικό. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει δηλαδή κανείς σε άλλο ε, συνεργείο για την πιστοποίηση και σε άλλο για την επισκευή. Μετά γίνεται μια παραπομπή στα ISO, ISO 1720. Και χωρίς να μιλάμε απαραίτητα για νομικό διαχωρισμό μεταξύ της ε, ε, επιθεώρησης και της επισκευής ή αποκατάστασης. Να μην φτάσουμε μέχρι το λεγόμενο unbundling. Με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να βρούμε μια λογική, πρακτική λύση. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση, πρόσθετη θα έλεγα, συμπληρωματική, για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα καταγράφονται τα σημαντικά κριτήρια και τα ορόσημα στη ζωή ενός ε, μηχανοκίνητου οχήματος. Είτε πρόκειται για τα χιλιόμετρα, είτε πρόκειται για τα ε, χρονικά σημεία της εξαγωγής των τεχνικών ελέγχων ε, ή άλλων επιθεωρήσεων, κυρία προβλήματα, κύρια ε, ανταλλακτικά που άλλαξαν, σημαντικά ανταλλακτικά που άλλαξαν κτλ. Θα όλα αυτά τα στοιχεία να ενσωματωθούν σε μια τεχνική βάση. Σε μια ε, βάση δεδομένων ώστε να μπορεί να, να ανατρέχει κανείς και να βρίσκει τα στοιχεία αυτά. Στη, στα τεχνικά παραρτήματα τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Σερατσάνη, ο οποίος αναλαμβάνει, η κυρία Σερατσάνη, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα στην Ιταλία και τη συγχαίρουμε εμένα, αλλά ε, ασφαλώς θα λάβουμε υπόψη τις προτάσεις της. Κύριος Λιμπεράτσκι. Αναφέρεται στα, στους φανούς φωτισμούς, στο σύστημα πέδησης, ε, στους καθρέφτες, επίσης κανόνες ε, κανόνες πιστοποίησης της καταλληλότητας για τα συστήματα παίδησης έχει προτείνει ο κύριος Σίμψον. Πάλι στους φανούς υπάρχει μια παρατήρηση, αλλά πάντως για, τις, ε, για την οικολογική διάσταση, είτε πρόκειται για το διοξείδιο του άνθρακα, είτε πρόκειται για τα οξύδια του αζότου ή άλλες ε, επιβλαβείς ουσίες, πρέπει μέσα στην ε, πιστοποίηση στην επιθεώρηση αυτή να αποφασίσουμε αν θα περιλαμβάνονται και αυτά τα στοιχεία των εκπομπών ή όχι, αν απλώς θα γίνεται χωριστά δηλαδή η διαπίστωση της ε, ρηπογόνου δράσης. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ τους αδέλφους για τη συνεργασία και περιμένω να ακούσω τη συζήτηση. Η κυρία Σενάλοβα είναι η επόμενη. Για το δεύτερο τμήμα που είναι οι επιθεωρήσεις, ο δικός τεχνικός έλεγχος δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέρφους για τα σχόλιά τους και για τα επικοδομητικά μάλιστα σχόλια τα οποία βελτιώνουν το κείμενο. Θέλω όμως να κάνω κάποια σχόλια, επιτρέψτε μου, στα κύρια σημεία που περιλαμβάνουν οι τροπολογίες που είναι 173 στο σύνολο του πακέτου. Όσον αφορά τη νομική μορφή, ορισμένοι συναδελφοί προτείνουν οδηγία αντί για κανονισμό. Και ο κύριος Φέρμπεθ και ο Μαρκίτσεβετς και άλλοι έχουν υποβάλει πολλές τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν την οδηγία. Πολλές φορές δεν είναι ολοκληρωμένη ενσωμάτωση στην νομοθεσία. Οπότε γι' αυτό εγώ λέω ότι προτιμώ ένα κανονισμό και μια που πρόκειται για πακέτο θα συζητάμε να συζητούμε αυτό το θέμα με τους συναδέλφους. Για μένα μια από τις κύριες προτεραιότητες είναι μια εισαγωγή βήμα-βήμα του συστήματος αυτού οδικού τεχνικού ελέγχου. Άλλοι συνάδελφοι δεν θέλουν αυτό το σύστημα. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να στηρίξω κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύω ότι το σύστημα αυτό αποτελεί μία από τις κύριες προστιθόμενες αξίες της πρότασης. Προκειμένου και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να διατηρήσουν τον, ε, τα φορτηγά τους, τα οχήματά τους σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν τροπολογίες 77, 78, 79 και πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ, διότι πιστεύω ότι οι, επι... οι επιθεωρήσεις που γίνονται στο δρόμο δεν οδηγούν στο σωστό αποτέλεσμα. Οι τροπολογίες 146-147 είναι επίσης τροπολογίες με τις οποίες δεν συμφωνώ, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα οδηγούσε σε διακρίσεις μεταξύ των χωρών μελών. Υπάρχουν όμως και άλλες τροπολογίες όπως αυτές που έχουν υποβάλει η κυρία Μπερμαν και η Γιάνσεν η 93 και 148 που προτείνουν μια περίοδο μάλλον εναρμόνισης δοκιμαστικά πριν να ε, τεθεί οριστικά το σύστημα προς εφαρμογή. Εδώ χρειάζονται παρετέρω διαβουλεύσεις. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι που καλύπτεται από τροπολογίες είναι το πώς θα διασφαλίσετε το φορτίο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες για μας. Ε, κύριοι Κόλεγεν και Ρίσπεθ έχουν την τροπολογία Τρία που εγώ δεν θα μπορούσα να δεχτώ, γιατί αυτό που προτείνει είναι μη οι υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε την εναρμόνιση των κανόνων που ελέγχουν το πόσο καλά ασφαλισμένο είναι το φορτίο πάνω στα φορτηγά. Να δούνε το βάρος τους, αν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η ελάχιστη εναρμόνιση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει όντως να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και θα ήμουν υπέρ του 5% για πάνω από 3,5 τόνους που πιστεύω ότι είναι το πιο ρεαλιστικό. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε πάντως το θέμα αυτό όπως επίσης και το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Η τροπολογία 83,5% όσον αφορά τα οχήματα τα οποία είναι καταχωρημένα, καταχωρημένα σε μια χώρα. Άλλοι προτείνουν 1%, άλλοι προτείνουν 3%. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε παρετέρω. Άλλες τροπολογίες τώρα από διάφορες πολιτικές ομάδες έχουν να κάνουν με το πεδίο εφαρμογής και αν θα συμπεριληφθούν και τα φορτηγά τύπου TAF5. Εγώ εδώ συμφωνώ με την τροπολογία 51 του κ. Σίμψον. Αλλά όπως έχω ήδη πει, οι τροπολογίες που δεν θέλουν να συμπεριληφθούν τα εμπορικά οχήματα και θερμοκούμενα κάτω από 3,5 τόνους είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε παρετέρω. Για μένα ότι ακόμα και τα μικρότερα οχήματα κάτω από 3,5 τόνων αποτελούν αυξανόμενο μάλιστα κίνδυνο για την οδική ασφάλεια και γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει να υποβάλλονται και αυτά στο σύστημα ελέγχων που προτείνουμε. Η τροπολογια 54, 63, Δεφέμπερ, Foster, Νταντέν, Ρικαμάσκε και βορτμαν Κόλ. Υπάρχει και ένας άλλος τομέας που καλύπτουν οι τροπολογίες και αυτός είναι ο ορισμός και η αλλαγή στον ορισμό. Πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο ορισμό όπως είπε και ο κύριος Κούν και αυτό πρέπει να συζητηθεί παρετέρω και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα καταλήξουμε τελικά σε έναν ορισμό αποδεκτό από όλους που θα είναι σαφής και που θα συνεισφέρει σε μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος χωρίς να αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες και αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι σημαντικό επίσης να δούμε το θέμα των, της ανεξαρτησίας των ελέγχων. Η κυρία Φώστερ έχει την τροπολογία τη σχετική, η οποία νομίζω ότι είναι προβληματική. Δεν θα πρέπει να είναι ο ίδιος που κάνει τους ε, ελέγχους τους τεχνικούς ε, στα κέντρα ελέγχου να κάνει και τους ελέγχους στο δρόμο. Η κυρία Λίσμπεθ, για παράδειγμα, έχει άλλη τροπολογία που αντιβαίνει στην πρόταση της Επιτροπής που μιλάει για τα 10 χιλιόμετρα απόσταση ανάμεσα στο σημείο που γίνεται ο έλεγχος και εκεί που γίνονται οι πιο λεπτομερείς έλεγχοι. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό λαμβάνοντας υπόψη και τις γεωγραφικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μελών. Τέλος, ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους τους συναδέρφους για την συμμετοχή τους στην συζήτηση για αυτό το τόσο τεχνικό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε. Και κυρία Σάβησα για τα έγγραφη κυκλοφορία οχημάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μια οδηγία που τροποποιεί τα έγγραφη κυκλοφορία οχημάτων είναι εκφύσεως ε, το μικρότερο από τα τρία έγγραφα που εξετάζουμε σήμερα και έγινε και λιγότερες ε, αναλόγως οι τροπολογίες. Δεν θέλω να μπω και να συζητήσω την πρόταση της Κομισιόν, την έχουμε ξαναζητήσει, θα πάω στους τροπολογίες κατευθείαν, τροπολογία 9, όπου ουσιαστικά αλλάζει μόνο η διατύπωση, ουσιαστικά την υποστηρίζω. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται, αλλά έχει μεταφράσει το κείμενο από τα αγγλικά στα εστονικά λανθασμένα. Και αν το επίσημο έγγραφο είναι το εστονικό, θα πρέπει παρακαλώ να το ελέγξουμε για να μην υπάρχουν προβλήματα. Τροπολογίες 10 και 11. Αφορούν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Συμφωνώ ουσιαστικά. Αυτό που δεν ε, συμφωνεί είναι η τροπολογία 12 του κυρίου Πάτπεν. Γιατί είναι σημαντική η προκειμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καλύψουμε όλα τα σημεία του πακέτου αξιο... οδικής αξιοπιστίας Είναι πολύ σημαντικό να μην επιτρέπουμε στους δρόμους οχήματα που δεν έχουν ελεγχθεί τεχνικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απαγορευτούν πλήρως. Αν δηλαδή το τεστ οδικής αξιοπιστίας έχει γίνει α, και το περάσουν τον έλεγχο, θα πρέπει να τους τη δυνατότητα να ξανακυκλοφορήσουν χωρίς να πρέπει να πούν ξανά σε ε, του ε, οχήματος. Κάτι που δεν επιτρέπει η τροπολογία του συναδέλφου. Εκτός αν εγώ δεν κατάλαβα καλά να νομίζω θα εξηγήσει καλύτερα μόνο στο τι εννοούσε. Δεν μπορεί να ούτε την 13. Και πάλι, ε, η ίδια αρχή, δηλαδή ε, η απόσυρση από το Μητρό, να ξεκινήσει δηλαδή την αρχή όλη διαδικασία, διαφωνούμε. Τροπολογία 14. Εδώ νομίζω πρέπει να υπάρχει κάποια παρανόηση και θα πρέπει συμπλοκή σε να το δούμε αυτό. Η νομική μας υπηρεσία θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά πόσο πρέπει να μιλήσουμε για ανάκληση ή παρακράτηση του πιστοποιητικού. ποιο είναι ο πιο όρο. Το 15 και 16. Ουσιαστικά ταυτίζονται με την δική μου τροπολογία 3. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική διατύπωση και για τις τρεις τροπολογίες τροπολογία 16, την οποία υποστηρίζω. Λοιπόν, ε, στο παράρτημα 1, σημείο 5. Παραπέμπει εδώ. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα. Τροπολογία 18 Πέρφερ ε, δεν την υποστήριζε για τους ίδιους λόγους. Τροπολογία 19. Για πιο ακριβή διατύπωση συμφωνώ. Τροπολογίες 20 και 21 επί της αρχής δεν διαφωνώ. Δίνουν πολλές νέες πληροφορίες στο κείμενο, κάτι που καθιστά το κείμενο πιο δυσανάγνωστο. Τροπολογία 22 της κυρίας Δεκάου Ταυτίστε με τροπολογία 5, τη δικιά μου. Τροπολογία 23 και πάλι τροπολογία 10. Επί της αρχής συμφωνώ. Αμφιβάλλω όμως κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να τηρήσουν αυτή την προθεσμία του 2016. Επίσης δεν συμφωνώ με τροπολογία 24. για το μέγεθος α7 που θα πρέπει να έχουν τα πιστοποιητικά. Δεν ξέρω κατά πόσο σε ένα μικρότερο μορφότυπο, κατά πόσον θα, θα, θα μπορούν να μπουν όλες τις πληροφορίες. Εγώ έχω εστονική εμπειρία. Στο μικρό αυτό πιστοποιητικό που έχουμε στα εστονικά έγγραφα υπάρχει αρκετός χώρος. 25 είναι ίδια με τη δικιά μου. Ε, νομίζω ότι μπορούμε εδώ να βρούμε μια κοινή διατύπωση. Αυτά από πλευρά μου και ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που ε, υπέβαλαν τροπολογίε που διευκρινίζουν το κείμενο. Έχουμε κάποια πράγματα να συζητήσουμε ακόμα με τον κύριο Μπράντμπαν, κατά τα λοιπά. Νομίζω ότι και εγώ και οι σκιώδες έχουμε συμφωνήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα σα αναφέρω το κατάλογο των ομιλητών και ποιο θέλει να προσταθεί, παρακαλώ.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 Εντάξει, μην φωνάξουμε τις ε, ιατρικές υπηρεσίες, ε. Όλα καλά. Ο κύριος Γρός πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα αναφερθώ εγώ σε κάποια γενικά θέματα της εκθέσεως. Επιμέρους ζητήματα θα αναφερθούν άλλοι συνάδελφοι σε σχέση με την έκθεση Κούν. η νομοθεσία νομίζω έχει να κάνει με την καθημερινή ζωή των πολιτών μας και γι' αυτό έχουμε καθήκον να εξηγήσουμε τι προσφέρουμε με την αυτή νομοθεσία και όχι να περιπλέξουμε την κατάσταση και την εικόνα για τους πολίτες με σε νέους λαβυρίνθους. Ε, πάντως οι προτάσεις δεν προς τη σωστή κατεύθυνση. αυτό το έγγραφο ταυτότητας θα λέγαμε για το κάθε όχημο το οποίο θα δίνει στοιχεία για, τις, για τα διανυθέντα χιλιόμετρα αλλά και πληροφορίες για μεγάλα ε, σχετικά ε, προβλήματα ή ατυχήματα που ενδεχομένω έχει περάσει το αυτοκίνητο αυτό έχει σημασία και δεν ξέρω γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό και σαν έγγραφο που εξυπηρετεί την ε, ε, συναλλαγή όταν πρόκειται να απολυθεί ένα αυτοκίνητο. Θα ήταν χρήσιμο, επιβάρυνση τέτοια διοικητική δεν προκύπτει και έτσι ε, είναι πολύ πιο ευχερής και ο τεχνικός έλεγχος η περιοδικότητα των ελέγχων. Όταν γυρνάει κανείς χρειάζεται πιο συχνά να επαληθεύει την κατάσταση υγείας του. Αυτό ισχύει και για τα οχήματα, εν πάση περιπτώσει, είτε σε ορισμένο χρονικό διάστημα, είτε μετά από ορισμένα χιλιόμετρα, 160.000 ε, είπατε, πρέπει να γίνεται ο τεχνικός έλεγχος. Αλλά πρέπει να γίνεται πάντοτε, ανάλογα με το τι θα αποφασίσουμε, και να μην λησμονούμε και τον υπερσυνοριακό ενδεχομένω χαρακτήρα και εδώ επανέρχομαι στο λεγόμενο car ότι δηλαδή στο διαβατήριο αυτών των αυτοκινήτων, όταν πάει να πουλήσει κανείς το όχημα του ε, πέραν των συνόρων, θα είναι χρήσιμο αυτό το διαβατήριο και ταυτόχρονα προς το συμφέρον της ασφάλειας των πολιτών του το κάθε κράτος θα έχει τη δυνατότητα να στήσει και επιπλέον ελέγχους. Για το συνεργείο επισκευών είχα κάνει μια πρόταση Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο τις παραδόσεις που έχουν επικρατήσει, αλλά να διδαχθούμε και από τις ε, θετικές εμπειρίες, εμπειρίες ε, σε διάφορα κράτη, όπου είναι ενιαίο το κέντρο πιστοποίησης και επισκευής. Θα μπορούσαμε να απαιτούμε μια ελάχιστη ε, ποιότητα ή μέγιστη ποιότητα, αναλόγως, αλλά πάντως σαφές είναι ότι όπου γίνεται η επισκευή θα πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα και ότι εάν κάποιος ε, κάνει παρατυπίες ή δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, θα κινδυνεύει να χάσει και τη δουλειά του και άρα θα είναι πολύ πιο προσεκτικός κανείς όταν ξέρει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Σέρλ Καντραβέ, θα μιλήσω αγγλικά επειδή επικεντρώνομαι στην έκθεση του κυρίου Κουν περισσότερο. Κάπως σύντομα. Μας ικανοποιεί πολύ η έκθεση του κυρίου Κουν, γιατί μας καλύπτει σε πολλά σημεία. Πρώτα απ' όλα το θέμα της εναρμόνισης των ε, τεχνικών ε, οχημάτων. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει πολύ καλά. Υπάρχει επίσης το ότι συμφωνείτε για το ότι οι χώρες που έχουν υψηλές προδιαγραφές δεν πρέπει να μειώσουν τις προδιαγραφές τους. Στηρίζουμε επίσης την άποψή σας για το ότι πρέπει να είναι κανονισμός και όχι οδηγία. Όσον αφορά τώρα τις ε, δοκιμές και το χρονοδιάγραμμα, ε, εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων, πάντως η βασική θέση μας είναι ότι εμεί θέλουμε το 4 1 1 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τις μοτοσυκλέτες εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να καλυφθούν από την πρόταση. Αλλά ίσως πρέπει να δούμε την τροπολογία της Μπενατέτ Βερνιό που λέει ότι μόνο τα δίτροχα και τρίτροχα πάνω το, από τέσσερα χρόνια θα πρέπει να ελέγχονται. Για τα τρέιλερς, εντάξει, φωνούμε και εμείς ότι δεν χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και ότι θα ήταν μεγάλη γραφειοκρατία και μεγάλο το κόστος αν τα συμπεριλαμβάναμε εδώ, τα ελαφρά ρημολκούμενα. Όσον αφορά τον ε, ορισμό του ποιο όχημα είναι κατάλληλο για το δρόμο, πρέπει να δείτε την έκθεση της Όλγας. Όσον αφορά τώρα τα γεωργικά οχήματα, που δεν πάνε πάνω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ έχουμε πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο πρέπει να συμπεριληφθεί η κατηγορία αυτή. Εμείς θα προτιμούσαμε να μείνει εκτός. Εκτός βέβαια από τα γεωργικά κίνα οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται στις ε, οδούς συχνά ή τα, για εμπορικού λόγους Τα κράτη-μέλη πάντως θα έπρεπε να μπορούν να πάνε πέρα από τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον το επιθυμούν. Όσον αφορά τέλος τα ιστορικά οχήματα, συμφωνούμε με την προσέγγιση του εισηγητή και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρούμε ένα καλό ορισμό για το τι ακριβώς είναι ένα όχημα ιστορικού χαρακτήρα. Τα συλλεκτικά οχήματα βασικά. συμφωνώ και με τις τροπολογίες Ματιέ ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις απάτες που επιχειρούνται. Ιδιαίτερα σε διασυνοριακές συναλλαγές καλό είναι να υπάρχει κάποιο είδος ταξινόμησης Είναι αλήθεια ότι η ιστορία ενός οχήματο είναι πιο δύσκολο να ανοιχνευτεί εφόσον πρόκειται για εισαγόμενο όχημα. Οπότε τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε όλες οι μετρήσεις να είναι πραγματικές αυτές που βρίσκουμε πάνω σε ένα όχημα. Πρέπει και αυτό να μπει στην έκθεση κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Κύριος Ευχαριστώ πολύ. Την τελευταία φορά που συζητήσαμε το θέμα αυτό, το μήλον της έρηδος ή το κυρίως το ζήτημα της διάρθρωσης των ε, κέντρων ελέγχου και των συνεργείων επισκευή σε σχέση με τους περιοδικούς ελέγχους. Εμείς είχαμε πει ότι δεν δεχόμαστε μία λύση ομοιόμορφη για τους πάντες. Ο κύριος Κούν φαίνεται να βρίσκει εναλλακτικέ λύσεις και δυνατότητα συμβασμού. Θα πρέπει να δούμε όμως τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Ε, ευχαριστούμε τον κύριο Γκρο για τις παρατηρήσεις του, είναι ευπρόσδεκτες. Κάποιες από τις χώρες με ε, ενοποιημένα συστήματα πρέπει να επισημάνουμε έχουν και τις καλύτερες επιδόσεις. Ενώ άλλες χώρες με χωριστά συστήματα σημειώνουν μείωση των προδιαγραφών εν ώψη της μείωσης και των τιμών, εν ώψη ενός ανταγωνισμού στις τιμές δηλαδή, περιορίζεται ε, και η προσοχή στην ε, τεχνική επάρκεια. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Βεβαίω είναι πολύ πιο εύκολο όταν κάποιο μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του και ε, για μισή μέρα ακόμη, για κανένα δύο ώρες σε ένα συνεργείο και να το πάρει έτοιμο και με την πιστοποίησή του. Είναι ένα σύστημα το οποίο και λειτουργεί καλά και αποτελέσματα φέρνει και διευκολύνει τον χρήστη. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος μπορεί να έχει συνηθίσει το σύστημα των δύο χωριστών κατηγοριών, μπορεί κάποιος άλλος να έχει συνηθίσει το ενοποιημένο, δεν χρειάζεται ο ένας να προσπαθήσει να πιέσει τον άλλον στην αποδοχή ε, του δικού του συστήματος. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της πρότασης χωρούν και τα δύο συστήματα. Για τα ρημουλκούμενα. Δεν νομίζω ότι το ρημουλκούμενα 0102 πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής. Βεβαίως ε, θα πρέπει και η υπερφόρτωση και η υπερβαστούριοτοχήτητος και η ανικανότητα στην οδήγηση να υπολογιστούν αλλά δεν υπάρχει λόγος ε, να σκεφτούμε ότι τα μικρότερα ρημουλκούμενα έχουν κάποια ιδιαίτερη, κάποιο ιδιαίτερο λόγο να υπαθούν. Θα συμφωνήσω επίσης με τον κύριο Αλκαντράουι για τα ε, οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στους δρόμους και τις εμπορικές χρήσεις. Για, τη ε, για το χιλιομετρικό κριτήριο πρέπει να επισημάνω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, αλλά ήταν ανέκαθεν, δεν έγινε τώρα τελευταία, διότι με περιορισμένη επιβάρυνση και με λίγη γραφειοκρατία θα μπορούσαμε να το λύσουμε, πιστεύω. Δεν υπάρχει λόγος να το διωγγώνουμε. Περιθώριο υπάρχει για τα ε, εξκαφικά, για τα ρημουλκούμενα, για τα ιστορικού ενδιαφέροντος οχήματα και περιμένω τις συζητήσεις στις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τζιχά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω να κάνω πρώτα κάποιες παρατηρήσεις για την έκθεση Κούν όσον αφορά τις δοκιμές. Εμείς υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες και θα τις συνοψίσω. Επιμένουμε να μην μειωθούν οι φιλοδοξίες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή περί το, το κάθε κάθε χρόνο. Μετά τα 165.000 χιλιόμετρα κάθε χρόνο να γίνονται έλεγχοι. Και μάλιστα εμείς λέμε αντί και 160 να είναι 120.000. Δεύτερο, δεύτερη ιδέα. Αυτό που μόλις ακούσαμε για αυτούς που επισκευάζουν τα αυτοκίνητα και για αυτούς που κάνουν τους ελέγχους. Εμείς έχουμε μια συμβαστική πρόταση για να καλύψουμε και αυτούς που οργανώνονται στα συνεργεία και αυτούς που, τους ελέγχους που γίνονται αλλού. Να μην υπάρχουν απαραίτητα διαφορετικά δίκτυα, αλλά να μην χρησιμοποιούνται τα ίδια κέντρα μέσα στον ίδιο χρόνο για το ίδιο όχημα. Δηλαδή να μην είναι το συνεργείο και αυτός που ελέγχει το όχημα ο ίδιος μέσα στον ίδιο χρόνο για το ίδιο όχημα. Είναι ένας συμβιβασμό που ίσως να σας βρει σύμφωνος. Τρίτον, άλλη μας τροπολογία είναι τα οξύδια του αζότου και τα σωματίδια και αυτά πρέπει να ελέγχονται στα οχήματα. Για την έκθεση ένα τώρα. Όλες μας οι τροπολογίες έχουν σαν στόχο να γίνονται οι έλεγχοι και για την ηχορύπανση, όχι μόνο για τις υπογόνες ουσίες. Αν βάλουμε λοιπόν κάποια ποσοστά, να μην ε, γίνει σε βάρος των ελέγχων που γίνονται στους δρόμους ε, για τους ταχογράφους, για τα φορτία των φορτηγών κτλ. Όχι επειδή θα έχουμε δηλαδή τους άλλους ελέγχους, να κόψουμε αυτούς τους ελέγχους, γιατί σε πολλές χώρες είναι τέτοια συνεργεία που κάνουν και το ένα και το άλλο. Μη μειωθούν οι έλεγχοι, για παράδειγμα, των ε, φορτηγών στους δρόμους. Αυτά είχα να πω για την έκθεση Κούν και την έκθεση Σελάνοβα. Αυτές είναι οι τροπολογίες που προτείνουμε και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβασμό. Ευχαριστούμε κύριε Ντουράν, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Φώστερ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για την έκθεση Κούν έχω κάποια σχόλια και μετά πολύ τα λόγια για την έκθεση Σενάλοβα. Δεν ε, θα αναφερθώ σε όλες τις τροπολογίες, στο όνομα του Θεού. Κάποια γενικά σχόλια. Δεν έχουμε αλλάξει θέση. Θεωρούμε ότι και δύο εκθέσεις, προεδρικός τεχνικός έλεγχος και ο ειδικός ε, έλεγχος και τα επαγγελματικές χρήσεις, ε, θα πρέπει ε, να είναι κανονισμό και όχι οδηγίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποια στοιχεία κλειδιά για του τόπου του δικολέχνου. Δεν έχουμε αλλάξει μα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εύρωστο στο σύστημα εν προκειμένου. Για εδώ και πολλά χρόνια 22.000 μικρέ επιχειρήσει και 50.000 επιθεωρητέ. Το να θεωρεί κανεί ότι αυτοί οι επιθεωρητέ, οι ελεγκτέ, επειδή επιθερούν επίπεδα, δεν ξέρω εγώ για τι πράγματα, ε, που είναι τόσο πολλά, δεν μπορούν να καταλήξουν σε ακριβή αποτελέσματα. Είναι ανόητο και γελίο αυτό. Κάνουν πραγματικά ενδελεχή έλεγχο και οι υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτά τα κέντρα είναι ε, αξιόπιστοι και ειλικρινεί, ε, και γι' αυτό και έχουμε αξιοπιστία στους δρόμους μας ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Αν τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα κράτη-μέλη θέλουν να έχουν διαφορετικό σύστημα, δικαίωμά τους είναι. Γι' αυτό Γι' αυτό θέλουμε ένα βαθμό επικουρικότητα και να έχουμε οδηγεί και κανονισμό προκειμένου. Τώρα για τα ιστορικά αυτοκίνητα, χαίρομαι γιατί λαμβάνονται και αυτά υπόψη, γιατί και αυτά πρέπει να λυθούν υπόψη και επιτατίθεται και το θέμα τη ανάκληση τη ε, ταξινόμηση οχημάτων. Με τον Τίβελ έχουμε πολύ καλό σύστημα ε, στη χώρα μα και είναι ένα ε, εύχριστο σύστημα, δεν είναι πολύ γραφειοκρατικό. Τι σημαίνει ότι ένα όχημα ε, απαγορεύεται στους δρόμους για λίγο χρόνο μπορεί να ξαναεπιστρέψει χωρίς πολλά προβλήματα. Δεν θέλουμε ούτε αυτό το σύστημα να το αλλάξουμε, γιατί λειτουργεί πάρα πολύ καλά με ταξινόμηση. Είναι ένα καλό ε, δρομένο σύστημα. Τώρα από εκεί και πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ένα άλλο καλό σύστημα στη χώρα σας, πολύ καλά κάνετε και εμείς το δεχόμαστε. Δεν συμφωνούμε με τις πράξεις και τις σχετικέ τροπολογίες ε, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε πλήρη έλεγχο για κάποια μέρους ε, σημεία και δεν θα πρέπει να υπάρξει εξουσιοδότηση προκειμένου στην Επιτροπή. Αυτά είναι τα σημεία κλειδιά. Έχουμε και α, Κάποιες προτάσεις ακούστηκαν για την άμεση πρόταση. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ουδέτεροι ε, προκειμένου. Αυτά είναι τα βασικά θέματα για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ε, λίγα λόγια αν με, μου επιτρέπετε, επειδή έχω το λόγο, λίγη ησυχία, για τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματική χρήση. Ε, παραλαμβάνω και εδώ θέλουμε οδηγία και όχι κανονισμό. Οι ε, συνάδελφοι, ήδη ανέφεραν κάποια σχόλια που να κάνω και εγώ, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Αυτό θα μα ανησυχούσε τα μάλλα. Γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι επιθεωρητέ μα κάνουν επιθεώρηση και έλεγχο πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογή αν δείτε επίση κατρεμουλκούμενα. Και αυτά θα πρέπει να ελέγχονται σε κάθε περίπτωση εφόσον είναι ελέγχος του βασικού οχήματο. Κάποιες άλλες μικρές λεπτομέρειες ε, τώρα. Εδώ συμφωνώ με όσο είπαν οι συνάδελφοι ε, για όσο είπαν να φύγουν από το σπίτι εφαρμογή για κάποια μικρά οχήματα. Συμφωνώ με το θέμα της οδικής αξιοπιστίας είναι ότι υπάρχουν και οχήματα που έχουν όλα τα πιστοποιητικά μαζί τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει α, ότι μας δίνει 100% αποτελέσματα. Θα πρέπει να λάβει υπόψη κανείς και ότι την ασφάλεια των, ε, των εγγράφων και θα πρέπει να δίνουμε την διακριτική ευχαίρεια ώστε να διατηρούνται σε ένα ασφαλές μέρος. Έπειτα, το σύστημα που έχουν στο Ηνωμένο προκειμένου είναι πάρα πολύ καλό και δεν θέλουμε να αλλάξει, δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί. Από εκεί και πέρα ο εισηγητής ε, α το λάβει υπόψη για τα τρέιλερ τα είπα. Έπειτα, άλλοι περιορισμοί για τους ελεγκτές, πεδίο εφαρμογή και περιορισμούς ε, των καθηκόντων τους. Όχι, θεωρούμε ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά ελεγκτές, είναι ξεκάθαρα τα καθηκόντά τους, είναι ξεκάθαρο τι πρέπει και τι πρέπει να κάνουν. Εμείς ε, δεν θα τους πειράζαμε καθόλου τους ελεγκτές μας, αν μας ρωτάτε, και από εκεί πέρα το παράρτημα να φύγει. Θεωρούμε ότι είναι πολύ περίπλοκο για τους ελεγκτές μας. Και αυτά τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ όλους οι ηγητές της σκληρή δουλειά που έκαναν. Αυτά είναι τα σχόλια από πλευρά μου. you, Ευχαριστώ κύριο Σαρτού. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Κούν, ιδιαίτερος για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, στα δί τρίκυκλα μπορούμε νομίζω να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Από τις αντιστοιχές και μόνο βλέπουμε ότι είναι πολύ συχνά θύματα τροχαίων δυστυχημάτων οι οδηγοί τους για τα τρίκυκλα αλλά και για τα δικύκλα ανεξαρτήτως ε, του αν φτάνουν μέχρι τις 80 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 200 ε, πρέπει να ε, αναγνωρίσουμε ότι είναι επικίνδυνη η χρήση τους ανεξαρτήτως ταχύτητας. Για τα οχήματα ιστορικής σημασίας, καλή είναι η πρόταση αρκεί να μην αποτελέσει την κερκόπορτα από την οποία θα μπουν και τα οχήματα που δεν έχουν ιστορική αξία για να αποφύγουν τους ελέγχους. Ο ρυθμός 4-2-2 για τους τεχνικούς ελέγχους είναι σωστός. Τώρα και τα πιο αμφιλεγόμενα ή διαφιλονικούμενα ζητήματα, αποχωρισμό ή διαχωρισμό του ελέγχου από την ε, επισκευή, η αρχή Τις ομοιόμορφες λύσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν ομοιόμορφες λύσεις, ούτε καν ε, πρόσφορο. Η 17.020 ISO, προδιαγραφή αυτή λέει ότι μπορούν τα κράτη-μέλη στο τρίτο, στο τρίτο στάδιο, τύπος γάμα δηλαδή, να αποφασίσουν μόνα τους εάν θέλουν να έχουν την αρχή των, ε, του διπλού ελέγχου ε, ή του διαχωρισμού του ελέγχου από την επισκευή καλύτερα, ώστε να βλέπουν τέσσερα μάτια το αυτοκίνητο ή όχι. Πάνω απ' όλα όμως κυριε και κύριοι συνάδελφοι είναι πολύ σημαντικό να μην, υποβαθμιστεί, ε, να υποβαθμιστούν οι απαιτήσει σε δεξιότητες των ελεγκτών και επιθεωρητών των οχημάτων εξαιτία αυτή τη ρύθμιση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να δώσουμε προσοχή. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Έχω 11 ομιλητέ στην Επιτροπή, του τρει εισηγητέ. Και άρα θα σας παρακαλούσα να περιορίσετε μόνο σε κάποια καινούρια παρατήρηση, να μην επαναλαμβάνετε τα όσα έχουν ήδη ακουστεί. Ο κ. Κάντσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους τρεις εισηγητές τρεις προτάσεις από πλευράς μας, εκ των οποίων δύο είναι κανονισμοί και μία προτάση οδηγίας. Αν θέλουμε να τηρούμε την αρχή της επικορικότητας για αυτά τα θέματα, είναι απαραίτητο Ιδίω η πρόταση κανονισμού ε, για την οποία έχει κάνει εκθέση ο κ. Κούν, οπωσδήποτε θα πρέπει να πάρει τη μορφή της οδηγίας. Θεωρώ απαραίτητο και απαράβατο όρο αυτό, για να μπορούμε να σεβαστούμε συγκεκριμένους κανόνες και περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε ε, στα κράτη-μέλη. Δεύτερο σχόλιο που ε, αφορά και πάλι την έκθεση Κούν αφορά το σεβασμό και την ε, ανάγκη να προάγουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, με λίγα λόγια. Μάλλον, στα λόγια είμαστε πάντοτε υπέρ των μικρομεσαίων, αλλά στις πράξεις δεν το κάνουμε. Και αν δούμε και την ε, πρόταση αυτή, θα δούμε ότι ουσιαστικά πιο πολύ ε, ικανοποιούμε τα συμφέροντα μιας πολυεθνικής σε σχέση με την επιβίωση μιας μικροεπιχείρησης ενός μικρού γκαράζ ε, που επισκευάζει ε, αυτοκίνητα. Θεωρώ ότι ε, όταν μιλάμε για αυτό το unbundling, για την αποδέσμευση, και το λέγαμε στους δρόμους, δεν είχαμε το θάρρος να το κάνουμε. Και τώρα μας απασχολεί να το κάνουμε ε, για το κάθε μικρό επισκευαστικό ε, γκαράζ. Ε, εκεί θα κάνουμε την αποδέσμευση. Λοιπόν, αρχή της επικουρικότητας και τήρηση της βασικής μας αρχής που είναι η προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρος, η κυρία Κρίσπακ. Euh, euh, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε τέσσερα μόνο σημεία και να μην επαναλάβω τόσα έχουν πει άλλοι. Νωρίτερα είχα επιμείνει για το ότι οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις και τα κράτη να φροντίζουν οι έλεγχοι αυτοί να γίνονται χωρίς διακρίσεις ανάλογα με την εθνικότητα του οδηγού ή τη χώρα προέλευσης του οχήματος και βλέπω ότι συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση Σολάνοβα αυτό. Κάποιοι μάλιστα συνάδελφοι προτείνουν να είναι εθελοντική η ταξινόμηση αναβαθμό επικινδυνότητας γιατί οδηγεί σε διακρίσεις μια τέτοια ταξινόμηση και δύσκολα θα λειτουργήσει. Γιατί θα έπρεπε να ειναι εθελοντικη η ταξινομηση αναβαθμού επικινδυνοτητας γιατι διασυνδεδεμένες και δύσκολο θα λειτουργησει γιατι θα δεδομένων γι' αυτά. Κατά τα άλλα βλέπω ότι για ορισμένες εξαιρέσεις για κάτω από 500 κιλά ε, ζητούν την εξαίρεση οι συνάδελφοι. Άλλοι όχι. Πάντως μην ξεχνάμε ότι η Σύμβαση της Βιέννης για την οδική κυκλοφορία λέει κάτω από 500 ε, δεν πρέπει όντως να έχουν ε, αριθμό κυκλοφορίας. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε να γελιοποιηθούμε εμείς οι Ευρωπαίοι και να βρούμε ένα συμβασμό. Στη χώρα μου αναρωτιόμαστε για τους ελέγχους αυτούς που για πολλούς πολίτες φαίνονται εντελώ περίεργοι. Έπειτα, συμφωνώ με την τροπολογία 122 της κυρίας Ντουρόν και εγώ έχω μια αντίστοιχη τροπολογία που προτείνει να γίνονται έλεγχοι στη, όσον αφορά τη ρήπανση των οχημάτων και όσον αφορά το οξύδια του αζότου. Τέλος, και για να απαντήσω λιγάκι και στους συναδέρφους, δεν θα μπορούσα να στηρίξω την πρόταση που θέλει να εξαρτήσει την χρήση των κέντρων ελέγχου από την γυτνίαση. Και έχω την τροπολογία με 130 που λέει να μην αναφερόμαστε σε αριθμό χιλιόμετρων, αλλά απλώ να λέμε ότι ο έλεγχος θα πρέπει να μπορεί να γίνεται στο πιο κοντινό κέντρο ελέγχου. Αν βάλουμε συγκεκριμένο αριθμό χιλιόμετρων, δυσκολεύουμε πάρα πολλές χώρες και τη δικιά μου μεταξύ άλλων, των οποίων τα οικονομικά υποφέρουν, για... είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί αν θέλουμε να φτιάξουμε επιπλέον κέντρα ή να αποκτήσουμε μια κινητή ομάδα ελέγχου, αυτό θα κόστιζε τόσα πολλά που δεν θα ήταν ρεαλιστικό. Ελπίζω οι συμβαστικέ τροπολογίες να περιλαμβάνουν κάπως και το πνεύμα των όσων σας είπα και μη μου ρίξετε σφυράκι κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριο Μπράτμπορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα το σχολείο μου στην εκθέση της οποίας έχουν λάβει τη σκιώδη εισηγή στη χαρα... την καταχώρηση οχημάτων. Αλλά μια και πρόκειται για οδηγία και όχι κανονισμό. Θα συμφωνήσω ότι και οι τρεις προτάσεις θα έπρεπε να υπαχθούν σε μια δέσμη οδηγιών. Για την κυρία Σάβεζα και την προσέγγιση της ως προς τις μου. νομίζω ότι τις έχει παρερμηνεύσει. Εμείς πιστεύω δεν θα έπρεπε να καταστήσουμε τους κανονισμούς αυτούς πολύ δεσμευτικούς να υπαγορεύουν λύσεις και έτσι όταν ορίζουμε ένα συγκεκριμένο θέμα για την άρση, την απόσυρση του κανονισμού αυτό θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Όπως και εσείς, κύριε Πρόεδρε, ως Βρετανός, ξέρετε ότι υπάρχει ε, μια διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο της απόσυρσης ενός αυτοκινήτου όταν αποφασίζει κανείς να το αποσύρει από τους οδούς ο ιδιοκτήτης του, πώς θέλει το σχετικό έντυπο στις αρχές, καταχωρείται κτλ. Το ίδιο και για το τεχνικό έλεγχο. ισχύει για μια συγκεκριμένη περίοδο και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ένα όχημα στους δρόμους αν δεν διαθέτει σχετικό πιστοποιητικό. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα που φαίνεται να συνοστίζονται στην, ε, στο σύνολο αυτό των προτάσεων για τροπολογίε σχέση με την αρχική πρόταση είναι ακριβώς αυτή η ιδέα, δηλαδή του να καταστεί λιγότερο δεσμευτικός ο κανονισμός. Συμφωνώ και με τις τροπολογίες κυρία να πω, παρότι σε κάποιες έχω κάποιες επιφυλάξεις, ιδιαίτερος όμως εκεί όπου, εκεί όπου μπορεί να επιβάλλεται μια συγκεκριμένη επιλογή στα κράτη-μέλη, η επιλογή ίσως και επικοινωνίας με τους ε, εταίρους κράτη-μέλη. Όμως ότι αυτά θα πρέπει να επαφίενται στην ε, διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Και μην ξεχνάμε ότι οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως του πολιτικού τους χρώματος πάντοτε μεριμνούσαν για την οδική ασφάλεια. Άρα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα περισσότερο προώθησης εκείνου που είναι πιο αποφασισμένος ε, για μια μεταρρύθμιση παρά να πιέζουμε εκείνον ο οποίος ε, καθυστερεί. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις όπως την Συμφωνία για τα προσωπικά δεδομένα πτήσεων, επιβατών πτήσεων, ε, το PNR έχουμε την ε, ίδια στάση ακολουθήσει και είναι και το πιο ασφαλή σύστημα αυτό. Άρα μόνο δίνουμε μια όθηση σε αυτόν που θέλει να προχωρήσει περισσότερο. Και σε αυτό η συνάδελφος νομίζω θα αντιληφθεί ότι εκεί όπου έχει ε, κάνει πιο παρεμβατικές προτάσεις με τις τροπολογίες της τότε θα χρειαστεί να τις διαχωρίσω από το κείμενο. Αυτά είναι τα σχολεία μου. Θα θέλαμε μια πιο απρόσκοπτη καταχώρηση οχημάτων, ανεξαρτός του εάν έχουν διαβεί σύνορα ή όχι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πρέπει και να μετατρέψουμε το όλο σύστημα σε ένα άχρηστο σύνολο κανόνων. Ευχαριστώ κύριο Πίρκερ. Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στην έκθεση του κυρίου Κούν. Τον ευχαριστώ θερμά για την έκθεση αυτή. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω τους στόχους που εξυπηρετεί. Είναι η βελτίωση της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές. Οι στατιστικές μας λένε ότι οι τεχνικές ε, τα τεχνικά προβλήματα, οι αστοχίες είναι ε, υπεύθυνα για 10% των τροχαίων ατυχημάτων. Βεβαίω υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ελέγχου. Σημαντικό είναι η επαλήθευση να γίνεται ανεξάρτητα ε, από την τεχνική, από το εργαστήριο, από το συνεργείο που θα γίνει η ε, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη η πιστοποίηση του επάρκεια, τεχνική επάρκεια του αυτοκινήτου, ανεξάρτητο του που θα γίνει η επισκευή. Γιατί υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν χωριστό σύστημα ε, με διαφορετικό συνεργείο από το κέντρο τη ε, πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου, ενώ κάποια άλλα έχουν ενιαίο σύστημα. Εδώ πέρα σημασία έχει να υπάρχουν χαμηλά ποσοστά ατυχημάτων. Δηλαδή στην ε, Αυστρία που είναι ενιαίο το σύστημα έχουμε χαμηλό ποσοστό, 2% μόνο ε, ατυχημάτων διότι είναι απολύτως εξασφαλισμένη η ανεξαρτησία στη δουλειά του ελεγκτή και βέβαια επικρέμονται και πάρα πολύ σοβαρέ ποινέ εφόσον κανεί παραβεί το καθήκον του. Άρα λοιπόν θέλουμε να αποφύγουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα λειτουργεί σωστά και αυτό θα πρέπει, είναι ο κίνδυνο ε, που κινδυνεύουμε να επιφέρουμε εφόσον επιμείνουμε όλοι για ένα ενιαίο σύστημα. Εάν είναι έτσι λοιπόν, προτιμότερο είναι να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία της ε, της αρχής της, ε, του κέντρου ελέγχου πάνω απ' όλα. Και εδώ στις προτάσεις παριθμών 12 και 13 που γίνεται λόγος για διαχωρισμό είναι νομίζω όχι λογικό, όχι απαραίτητο, διότι και το σύστημα και συστήματα που λειτουργούν σε κάποια κράτη-μέλη διαταράσει και δεν βελτιώνει σε τίποτα την ε, ανεξαρτησία. Για δε προτάσεις ως προς τις ε, όπως ε, το προσορισμό προτύπων, προδιαγραφών. Σε αυτό δεν έχω εγώ αντίρρηση, μεν, αλλά εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει μέσα στις προδιαγραφές η ε, προϋπόθεση, παραδείγμα ότι μόνο κάποιος νομικός μπορεί να κάνει τον έλεγχο, μπορεί να πιστοποιεί τον έλεγχο, τότε δεν βλέπω ε, σε τι θα μπορούσε αυτό να εξυπηρετήσει. Έχουμε πολλές, ε, νομικό πρόσωπο να κάνει τον έλεγχο, τότε ε, δεν βλέπω σε τι αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει στην ε, Αυστρία. Έχουμε ένα 70 περίπου επιχειρήσεων που λειτουργούν και που εάν εισαχθεί αυτός ο όρος θα αποκλείονταν από τον τεχνικό έλεγχο. Δηλαδή έχουμε προτάσεις που είναι πολύ απόλυτες του διαχωρισμού ή του ε, προτύπου ή της ε, νομικής προσωπικότητας εν πάση περιπτώσει που μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και την πιστοποίηση οι οποίες δεν εξυπηρετούν την ασφάλεια. Η ασφάλεια θα εξυπηρετηθεί ε, και με το να διατηρηθούν συστήματα που λειτουργούν ικανοποιητικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Σκόχ. Ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ όλους τους εισηγητές. Θα ήθελα και στις δύο εκθέσεις να τοποθετηθώ. Καταρχά είμαι υπέρ της λύσης οδηγίας, γιατί έτσι μπορούν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω συστήματα ελέγχου, επαλήθευσης, πιστοποίησης. Δεύτερον, είμαι υπέρ του διαχωρισμού του ελεγκτή με την έννοια ότι όταν δύο ζευγάρια μάτια παρακολουθούν ένα όχημα είναι καλύτερο από το να το βλέπει μόνο ένα. Τρίτον, η πρόταση για 4 και 2, 2 χρόνια μετά για τον έλεγχο, για την ε, περιοδικότητα του ελέγχου, δεν με ενοχλεί, δεν με ανησυχεί, αλλά βέβαια βλέποντας ότι αυτοκίνητα τα οποία έχουν ηλικία 10 ετών δεν είναι απαραίτητα ε, πιο επικίνδυνα, προτείνω ε, μία λύση, γιατί εάν πούμε στους πολίτες ε, της Ευρώπης «Α, κοιτάξτε, εάν έχετε αυτοκίνητα πάνω από 10 ετών, μπορείτε να τα πηγαίνετε εσείς για έλεγχο, όποτε το θεωρείτε σκόπιμο ε, και κάθε χρόνο αν θέλετε», τότε θα δούμε ότι δεν θα αντιδράσει, δεν θα αποκριθεί ο κόσμος, γιατί θα σκεφτεί τα έξοδα και τελεπορία κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε άλλες λύσεις. Για, τον, για το ταχόμετρο και το το κίνδυνο να είναι πειραγμένο και να διορθώνεται τα χιλιόμετρα που έχει δίνει στο αυτοκίνητο. Πρέπει αποτελεσματικά να το καταπολεμήσουμε. Επίσης, για την κυρία Σαβισάρ, έχω μια ερώτηση. Το θέμα της ασφάλισης δεν ξέρω πώς θα καλυφθεί. Όταν ε, επιστρέφονται οι πινακίδες ενός αυτοκινήτου, δεν ε, σβήνει και κάθε είδους ε, ευθύνη ε, από, νομική ευθύνη δηλαδή από το αυτοκίνητο αυτό. Δεν πάβουμε δηλαδή να είμαστε υπεύθυνοι για κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ή να προκαλέσει το αυτοκίνητο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα της ασφάλισης. Φέρμπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομο ω σκιώδη ηγητής της ομάδας μου για την έκθεση της κυρίας Σενάλοβα. Λαμβάνω το λόγο. Αλλά θα πω και δύο λόγια για τον κύριο Κούνα θα μπορούσε για τα φορτηγά αυτοκίνητα να προβλέπεται μια τακτικότερη επαλήθευση της, των τεχνικών στοιχείων, τακτικότερη δηλαδή από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, σε θελοντική βάση, η οποία όμως θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί θετικά ε, υπέρ του ιδιοκτήτη. Και έτσι και ενθαρρύνουμε αυτόν ο οποίος θέλει να κάνει κάτι περισσότερο, να είναι πιο προσεκτικός και καταγράφουμε, πιστοποιούμε αυτήν την ε, αξιοσημείωτη συμπεριφορά. Κατά τα άλλα, για τα επιχειρήματα οδηγία ή κανονισμός, νομίζω ότι εκεί όπου υπάρχουν καλής ε, ποιότητας συνεργεία και με την αρχή το, να παρακολουθούν, να ελέγχουν το αυτοκίνητο δύο ζευγάρια μάτια, όπως είπε ο κ. Κόχ, έχουμε μια καλή λύση μπορούμε να την προαγάγουμε. Το σύστημα ε, αξιολόγησης κινδύνου με προβληματίζει πρέπει να πω. Ένα όχημα το οποίο ή ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλής επικινδυνότητας δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό για να είμαι ειλικρινή. Δεν γνωρίζω ακριβώς τεχνικά στοιχεία, αλλά δεν θα έπρεπε πάντα να είμαστε ω δυνατόν πιο καλοί. Εάν κάποιο χρησιμοποιείται ω ε, ενό κάποιου επίπεδου επικίνδυνοτης, θα πρέπει να γίνεται η απαλήθευση και η διόρθωσή του πιο τακτικά. Αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Στο άρθρο 5 για τα ξένα αυτοκίνητα θα υπάρχει μια ε, ποσόστοση ανάλογα με την ε, συμμετοχή τους φαντάζομαι με την συχνότητα εμφάνισής τους στις οδικές μεταφορές. Παραδείγματι Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία που έχουν πολύ μεγάλη συχνότητα ξένων αυτοκίνητων που κυκλοφορούν ε, θα έχουν πολύ πιο πολλούς ελέγχους από ότι τα κράτη της περιφέρειας που ε, βλέπουν λιγότερα ξένα οχήματα. Η κατάθεση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου ή αλλιώ ενό αντιγράφου, σε αυτό το ζήτημα εγώ θα προτιμούσα πάντα το πρωτότυπο, είναι πολύ πιο ασφαλέ. Επίσης, ε, στο, σημείο, στο άρθρο 5 που αναφέρεται η δυνατότητα για έναν οπτικό έλεγχο. Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί ήδη ένας πρώτος έλεγχος, μια πρώτη επιθεώρηση μπορεί να δώσει σαφής, ε, σαφή εικόνα για το αυτοκίνητο. Κύριε Σαβάνα. ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω και εγώ τη δικιά μου τη φωνή σε εκείνον οι οποίοι μίλησαν για οδηγία. Πρέπει να τηρηθεί εδώ η αρχή της επικουρικότητας. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω. Και δεν το άκουσα αρκετά. Γιατί άραγε. Οι πληροφορίες, τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε για τις μοτοσυκλέτες Και αυτό το λέω γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει έντονη επιθυμία να συμπεριληφθούν. Ίσως να είναι καλό, αλλά δεδομένου ότι δεν έχουμε τα δεδομένα, μήπως είναι καλύτερα να μην τα συμπεριλάβουμε. Έχω τις αμφιβολίες μου δηλαδή, αλλά τέλος πάντων μπορεί να είναι και λεπτομέρεια. Κατά τα άλλα είναι εξαίρετη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ τους συζητητές. Η κυρία Τικάο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τόσο έχουμε ήδη ακούσει, οι μοτοσυκλέτες πολύ συχνά εμπλέκονται σε ατυχήματα. Γι' αυτό και εγώ στηρίζω την ιδέα αυτή να γίνονται υποχρεωτικά έλεγχοι και στις μοτοσυκλέτες. Έχουμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Σαββισάρ. Εγώ είμαι σκιώδης η συγγήτρια από πλευράς των σοσιαλιστών και στηρίζουμε την αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων που γίνονται δηλαδή σε άλλες χώρες μέλη. Στηρίζουμε την ιδέα της εισαγωγής επίσης ηλεκτρονικών μητρών. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να πετύχει αυτό. Και είναι πολύ βασικό να υπάρχουν τέτοια εθνικά ή ηλεκτρονικά μητρώα που να συνδέονται μεταξύ των διαφόρων χωρών. Όσον αφορά τώρα την μορφή του πιστοποιητικού, εγώ δεν πιστεύω ότι αν ε, επιβάλλουμε μία νέα μορφή, όπως είδαμε σε κάποιες τροπολογίες, α6 ή κάποια άλλη μορφή, πώς θα γίνει η εναρμόνιση αν επιμείνουμε στο σημερινό, που είναι λιγότερο από α4, τότε μπορούμε να συμπεριλάβουμε και όλες τις άλλες πληροφορίες που θέλουμε. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες 13 και 15, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αλλάξει ο ορισμός αποσύροντας ή ακυρώνοντας το πιστοποιητικό αυτό. Πάντως η τρέχουσα οδηγία αναφέρει τις περιπτώσεις που μπορεί να γίνει αυτό. Θα ήθελα κατά τμήματα ψηφοφορία εκεί ή με τη βοήθεια των σχεδόν εισηγητών ή των εισηγητών. Ίσως καταφέρουμε πάντως να βρούμε ένα συμβασμό για το θέμα του ορισμού. Όσον αφορά τώρα τις εξαιρέσεις για την ακύρωση του πιστοποιητικού καταχώρησης για τα συλλεκτικά οχήματα σίγουρα μπορεί να επηρεάσουν την οδική ασφάλεια τα οχήματα αυτά, αν και δεν κυκλοφορούν τόσο πολύ όσο τα υπόλοιπα οχήματα. Αλλά να μην χρειάζεται νέα καταχώρηση. Στο 3α νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος, γιατί στο παράρτημα 1, σημείο 2, 4, εγώ δεν το βρίσκω. Ίσως πρέπει διμερώς να το συζητήσουμε για να δω κατά πόσο αυτό το στοιχείο υπάρχει κάπου, τέλο πάντων που θα έπρεπε να υπάρχει. Η έκθεση πιστεύω ότι είναι καλή και είμαι πεπισμένη ότι μετά την ψηφοφορία θα καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική θέση για όλους. Παρακαλώ τώρα, κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Είναι πολύ βασικό να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές και πληροφορίες μεταξύ μας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή η κατάσταση βέβαια από χώρα σε χώρα διαφέρει και γι' αυτό και επιμένω, όπως είπαν και άλλοι, ότι πρέπει να τηρούμε την αρχή της επικούρικότητα. Εξάλλου οι συζητήσει στο Συμβούλιο θα είναι πολύ πιο εύκολε γιατί σίγουρα δεν συμφωνούν με τον κανονισμό. Είναι ένα τομέα αυτό, καταλαβαίνετε, πολύ σοβαρός βέβαια. Έχει πολύ σημασία να υπάρχουν έλεγχοι ή οδικοί κώδικες που να ρυθμίζονται ευρωπαϊκά. Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με τα δίτροχα και τρίτροχα μηχανοκίνητα οχήματα. Όντως, τα δίκυκλα εμπλέκονται σε πολλά ατυχήματα, αλλά όχι εξαιτίας τεχνικών αστοχιών, κάτω από 1%. Δεν πρόκειται βέβαια να λύσουμε έτσι το θέμα των ατυχημάτων όπου εμπλέκονται δίκυκλα. Η πρότασή μου λοιπόν στον κύριο Κιούν είναι ναι, ναι, υπάρχουν χώρες όπου είναι υποχρεωτική έλεγχη αυτή, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες όπου ο κόσμος δεν θέλει να είναι υποχρεωτική αυτή η έλεγχη. Γι' αυτό και προτείνω στον εισηγητή να αφήσει στην επικουρικότητα αυτή την απόφαση, δηλαδή να αφήσει τις αρχές των κρατών μελών να αποφασίσουν. Γιατί, Γιατί αναγνωρίζουμε ότι αν ε, κάπου είναι υποχρεωτική έλεγχη, ε, τότε η οδηγοί των δικύκλων ξέρουν ότι για να κυκλοφορήσουν στις χώρες αυτές πρέπει να έχουν ε, τον έλεγχο. Είναι λοιπόν θέμα επικουρικότητας που πιστεύω να σεβαστούμε και αυτό είναι ο συμβασμός που προτείνω. Ο κύριος Λιμπεράσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αφαιρθώ στις ε, δύο αυτές πρώτες εκθέσεις, να ευχαριστήσω και τον κύριο Κούν και την κυρία Στενέλοβα για το έργο Σε ό,τι αφορά την έκθεση Κούν, είμαι ε, στην παράταξη εκείνων που θεωρούν ότι το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Οπότε, μην ξεχνάμε την υπάρχουσα πραγματικότητα. Εμείς στη χώρα μας έχουμε ένα χωριστό σύστημα ε, τέτοιων μικρών ε, συνεργείων και κέντρων τεχνικού ελέγχου και θα πρέπει να παραμείνει αυτό όσα έχει. Το σύστημα επίσης ελέγχου των καυσαερίων ε, πρέπει να παραμείνει όσα έχει. Εμεί ε, προβλέπουμε από τον έλεγχο καυσαερίων στο χώρο τεχνικού ελέγχου. Εδώ μιλάμε και θέσει εργασία, Αν αλλάξουμε το σύστημα αυτό, θα έχουμε απώλεια θέσεων εργασίας. Λίγα λόγια τώρα και για την έκθεση σε άλοβα. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες, την 92-44-37 εν παραδείγμα αναφέρω, γιατί το 5% ως ελάχιστο ποσοστό ελέγχου αντί για 3% ώστε με τον τρόπο να έχουμε προσδραστές εργασία στο τομέα του τεχνικού ελέγχου. 3% κατά τη γνώμη μου είναι εντάξει, λογικό ποσοστό. Αλλά γιατί να μην τον εμβάσουμε στο 5% αν μπορούμε, αν θέλουμε να ελέγξουμε μια εταιρεία με προφίλ υψηλού κινδύνου, τελικά θα καταλήξουμε σε ένα αυθαίρετο σύστημα. Ένα σύστημα δηλαδή όπου ο ελεγκτής αποφασίζει ποια εταιρεία θα ελέγξει ή όχι και έτσι άλλε επιχειρήσει θα τη χάνουν ελέγχου και κάποιες άλλες δεν θα ελέγχονται καθόλου. Θεωρώ ότι αυτή η λύση που προτείνεται είναι αρκετά επικίνδυνη. Δεν πρέπει λοιπόν να εισαχθούν αυτά τα μέτρα. θα πρέπει να δείξουμε να σαφές, μια σαφή στάση προκειμένο. Από που και προέρχονται προβληματικά οχήματα, αυτά θα πρέπει να ελέγχονται. Το έχω συζητήσει το θέμα και με τον κλάδο των μεταφορέων ε, και αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθείται σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο pattern συμπεριφορά, όταν υπάρχουν πινακίδε από μια συγκεκριμένη χώρα, σταματάτε το όχημα για έλεγχο κτλ. Αυτός είναι και ο φόβος πολλών ε, μεταφορέων ότι θα μπουν σε μια τέτοια επικίνδυνη κατηγορία και συνεχώς θα τους σταματούν για έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Τέλο, πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Επιτροπής και Θέλω να πω και εγώ λίγα λόγια και να αναφερθώ και στις δικές μου τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα για το θέμα των τροχών. Είναι ένα θέμα ε, που γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες. Το θέμα λοιπόν των πλημνών είναι πολύ σημαντικό, αλλά το γνωρίζετε δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες. Έπειτα, έχω και ένα άλλο πρόβλημα και θέλω να σας το πω. Μπορεί, επειδή προέρχομαι από μια χώρα που δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, όλοι αναγνωρίζουν την εξαρτησία των ελεγκτών. Ακόμα και αν οι ελεγκτές είναι αυτοί που έχουν επισκευάσει το αυτοκίνητό σου. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε αυτή την αναγκαστική διάκριση που πρέπει να γίνει σκεφτείτε και πόσο ε, επιπρόσθετο βάρος θα σημαίνει για κάποιες χώρες. Γιατί να μην αφήσουμε στη θέση του ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί μια χαρά. Δεν ξέρω πώς θα δικαιολογήσουμε τις επρόσθετες δαπάνες και το βάρος σε αυτά τα κέντρα ελέγχου που έως τώρα κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Φαντάζομαι όμως για να το προτείνετε κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα θα υπάρχει πρόβλημα εκτός από αυτά που είπε ο κύριος Μπέρκερ για να ε, εξαιρέσω την Αυστρία και τον Αμένο Βασίλειο, δεν καταλάβω τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες σε ό,τι αφορά τα τρακτέρ και τα τρέιλερ. Και εγώ είπα κάποιες τροπολογίες στην ε, έκθεση κυρία Σενέλοβα για να μπορέσουμε να βάλουμε μεν και αυτές τις κατηγορίες του πεντεφαρμογής χωρίς όμως να δημιουργούμε ε, πολύ ψηλές απαιτήσεις για τρέιλερ και τρακτέρ καθώς ε, συνεπάγονται πολύ χαμηλό κίνδυνο στους δρόμους. Ούτως ή άλλως οποιοδήποτε όχημα κινείται στους δρόμους θα πρέπει να, είναι, ε, να έχει ειδική αξιοπιστία. Σκεφτείτε τώρα να συμπεριλάβουμε και όλα τα αγροτικά οχήματα που βγαίνουν από το ένα χωράφι για να μπουν στο άλλο τι νόημα έχει. Για τα μικρά τρέιλερ, το 01 και 02 δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μπουν και αυτά ε, στο πεδίο εφαρμογή. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Ένα από τα προβλήματα κατά με είναι ότι έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθώντα λοιπόν να βρούμε τώρα τη μέση λύση, είναι κάτι που δεν λειτουργεί πάντοτε. Τελευταίο σχόλιο για ε, τα υγρά των φρένων ε, και τον ε, σχετικό τεχνικό έλεγχο. Μόνο ένα συνάδελφο ενδιαφέρεται συνεχώ για τα υγρά φρένων και πολύ ορθά μα είπε ότι αυτή η δοκιμή ουσιαστικά είναι δοκιμή για το περιεχόμενο των υγρών. Αλλά δεν είναι το κατάλληλο τεστ για τα υγρά φρένων. Ξέρετε εγώ που διαφωνώ με σας κύριε Φρέμπερ ότι λέτε κανένα τεστ για τα υγρά φρένων. Αν υπάρχουν όμως καλύτερα τεστ, όπως είναι ε, τα τεστ E, ε, για το σημείο βρασμού δηλαδή του υγρού των φρένων, ε, τότε αυτό το τεστ πρέπει να προκρίνουμε και όχι το τεστ περιεκτικότητας των υγρών. Γιατί στα υγρά των φρένων η περιεκτικότητα μας οδηγεί σε πολύ αναξιόπιστα αποτελέσματα και δίκιο έχετε που λέτε να καταργηθεί να τα πούμε μεταξύ μας, μπας και σας πίσω. Το σημείο βρασμού είναι το καλύτερο τεστ που μπορεί να γίνει για τα υγρά φρένων. Λοιπόν, αυτά είναι και τα δικά μου σχόλια. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλει και αυτός, να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ο κύριος Ονίλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον που εκφράσατε ε, για αυτή την πρόταση. Ε, η δυσκολία στο όλο θέμα είναι ότι συζητάμε για βελτιώσεις ε, και έχουμε μπροστά μας τρεις εκθέσεις εξαιρετικής ποιότητας. Ε, θέλω πραγματικά να επενέσω και τους τρεις εισηγητές, ε, οι οποίοι μας υπέβαλαν υπόψη μας πολύ εξαιρετικές εκθέσεις. Δεν δεν εννοώ ότι οι άλλε δεν είναι τόσο καλές, αλλά εν προκειμένου βλέποντα και την παρουσίαση που έκαναν ε, και για τον τρόπο τον οποίο βλέπω και τι αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε σε στο ίδιο μήκος ε, και εμείς. Λίγα πράγματα έχω να πω, λίγα στοιχεία που έθεσαν ε, πολλοί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Κατηγορία L και σε περίληψή τα δίτροχα και τα τρίτροχα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους περιοδικούς ελέγχους, είναι καθοριστική σημασία και για λόγους ε, συγκέντρωση υποδικών στοιχείων, αλλά και για να είμαστε ακόλουθοι με την τεχνική νομοθεσία που έχει θετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, σε ό,τι αφορά αυτή την κατηγορία οχημάτων. Μπορούμε να γνωρίσουμε βεβαίως μια κάποια ευελιξία, η οποία θα ήταν η εξή πιθανόν Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τις πιο σημαντικές κατηγορίες, δηλαδή κατηγορίες που ε, έχουν περίπλοκα συστήματα, όπως το σύστημα EBS. Υπ' αυτή την έννοια θα λέγαμε να συμπεριλάβουμε και άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με την πολύ πρόσφατη νομοθεσία ε, κρυμμένων ειδών, τύπων, συγγνώμη, τύπων, ώστε να υπάρχει απόλυτη συνάφεια και ε, αντιστοιχεία. Η ευελιξία πάλι. Η ευελιξία μπορεί να σημαίνει πολλά και μπορούμε σε πολλά σημεία να επιδείξουμε περαιτέρω ευελιξία. Συμφωνώ, Πρόεδρε, με αυτό που είπατε για τα τρέιλερ. Και εσεί και οι συνάδελφοί σα το είπαν. Ίσως να πρέπει να περιοριστούμε σε εκείνα τα τρέιλερ, σε εκείνα τα ερμουλκούμενα ε, τη κατηγορία 02 που ε, φέρουν κάποιο φορτίο συμπεριλαμβάνοντα και αυτά που έχουν και φρένα. Τώρα για τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στην Επιτροπή σας. Ας δούμε τα δεδομένα, ας δούμε τα στοιχεία. Έχουμε ισχυρά στοιχεία που μας δείχνουν ότι η ηλικία του οχήματος ε, συνδέεται άρρηκτα με τα τεχνικά προβλήματα που οδηγεί σε ατυχήματα. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να επισημάνω και πάλι πόσο σημαντικό είναι αυτή η πρόταση να χρησιμοποιηθεί για να επιτύχουμε την εναρμόνιση ε, των τεχνικών ελέγχων ε, που θα πρέπει να γίνεται ετησίω για οχήματα από μια ηλικία και πάνω. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται ε, σε κάποιους από εσάς πολύ προβληματικό, αλλά θέλω να σας πω ότι η επιστήμη, τα αποδεκτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τροχαία ατυχήματα, επισημαίνουν όλο και πιο συχνά το στοιχείο της αμοιβές αναγνώρισης όταν πάνω το 15% των οχημάτων σήμερα είναι οχήματα από δεύτερο χέρι, είναι πολύ λογικό λοιπόν, παράλληλα με την αμοιβαία αναγνώριση, να μπούμε σε περαιτέρω ε, εναρμόνιση και να μπαίνουν αυτά τα οχήματα σε αιτήσιο έλεγχο. Σας παρακαλώ, εν προκειμένου, μελετήστε καλά τις πολύ καλές τροπολογίες ε, των κυρίων Γκρός και για να βρούμε μια μέση οδό πώς να συνδέσουμε περισσότερο τον ετήσιο έλεγχο με αντικειμενικά κριτήρια όπως είναι τα χιλιόμετρα, χιλιάδε χιλιόμετρα και, χιλιάδες χιλιόμετρα και πάνω, αν έχουν τα λοιπά. Ενημερωτικά, ενημερωτική πλατφόρμα και βεβαίως και εμείς συμφωνούμε για την φύση των κέντρων ελέγχου βλέπουμε αρκετή κατανόηση αυτά που είπατε αρκετή και αυτό που η κυρία Φώστρη και ο κύριος Μπένιεν συγκεκριμένα. Ίσως υπάρχει όμως μια παρανόηση εδώ. Δεν θέλουμε εναρμόνιση για την φύση αυτών των κέντρων ελέγχου. Στην έκθεση Κούν δεν είδα πουθενά να λέγεται κάτι που να ξεπερνά, αν θέλετε, αυτό που και εγώ θα θεωρούσα θεμητό. Δηλαδή μια γενική αρχή που να λέει ότι αυτός που επισκευάζει το αυτοκίνητο, το όχημα, δεν είναι ο ίδιος που μετά θα κάνει τον έλεγχο και θα δώσει πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Ε, αυτή λοιπόν ε, η τροπολογία ε, του κύριου Κούν είναι θεμητή τροπολογία και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα σκαμμένα. Σε ό,τι αφορά την έκθεση της κυρίας Εναλόβα, Συμφωνώ με απόλυτα με όλες τις αρχές που επισημαίνει ιδιαίτερως. Τώρα μια σειρά τροπολογιών εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα και τις υποστηρίζουμε. Θέλουμε ελέγχου να διεξάγονται και εσείς πρόεδρε το είπατε και άλλοι της συναδελφοί σας Φιντάνσα Ντυρόν προτείνετε τροπολογίες ε, για να ε, γίνονται περαιτέρω έλεγχοι στους τροχούς, ε, στα λάστιχα κλπ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δείξουμε την ίδια ευελιξία και πάλι για τα ρημολικούμενα, για τα τρέλερ, να συμπεριλάβουμε μόνο τα ρημολικούμενα υψηλού αντικτύπου. Και όσο αφορά την απόσταση από τα κέντρα ε, ελέγχου, βλέπουμε αρκετή κατανόηση την πρότασή σας, δηλαδή ενδεχομένως να διαγράψουμε τον ακριβή αριθμό χιλιόμετρων από το κέντρο και να μιλήσουμε για το ε, κοντινότερο κέντρο ελέγχου έτσι θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτό το κανόνα πιο εύκολα σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα κυκλοφορία των οχημάτων, πολύ σημαντική πρόταση και αυτή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα με όλη τη δουλειά που έκανε ε, η κυρία Σαϊφσέρ στο, στο, στο κείμενό της, καθώς διευκρινίζει πολύ την πρόταση και μιλάει για θέματα όπως είναι το ε, μορφότυπο που θα πρέπει να έχει το έγγραφο, ε, κοινό μορφότυπο για να είναι εύληπτο το έγγραφο στον όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτέλους προτάσεις όπως ενίσχυση του καθεστώτος και για την ε, ε ταξινόμηση αλλά και για την διαγραφή από τα μητρώα των οχημάτων και προτάσεις που συνδέονται και μεταξύ το όχι, με στο τέλος της ζωής του ε, όταν αποσύρεται από την κυκλοφορία θα πρέπει να έχει και αυτόματη απόδειξη της διαγραφής του από τα αρχεία. Ε, θεωρώ ότι και εδώ όλε οι τροπολογίες που έχουν σκοπό μια καλύτερη και ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής και ιδίως την πλατφόρμα τα λέξη πληροφορία των των μελών είναι κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε και συνάδει και απόλυτα με μια σειρά τροπολογιών από τις Επιτροπές Ήτρα και Ήλκο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε οι συγητές. Πολύ σύντομα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Κύριε Κούν πρώτα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα πολλά σχόλια που έλαβα στην έκθεσή μου. Κάθομαι λοιπόν εδώ, ακούω και σοφός πιο πολύ δεν έγινε. Διότι αν παίρναμε την πρώτη συμφωνία του Συμβουλίου και ακούγαμε τι είδου θετικέ αναφορές ε, παρουσίασαν οι διάφοροι συνάδελφοι, τι συγκρίνουμε με τα κράτη-μέλη από τα οποία προέρχονται, θα είχαμε ακριβώς ταύτιση της εικόνας και στο θέμα των ατυχημάτων και στο θέμα των νεκρών και της εξοπιστίας των ελέγχων κτλ. Στον τεχνικό τομέα νομίζω υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Είναι καθοριστικά. Το αν θα είναι οδηγία ή κανονισμός έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό παρακαλώ και τους και ηγητές και τις πολιτικές ομάδες να προχωρήσουν στην επιλογή μίας γραμμής για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εάν εισάγουμε μια σειρά από εξαιρέσεις δεν αξίζει τίποτα ο κανονισμός. μπορούμε να πούμε ότι προχωρούμε στη λύση της οδηγίας, βγάζουμε τα παραρτήματα, ε, μιλάμε μόνο για το μέγεθος, ε, τα, τα, μεγαλύτερους, τα μεγαλύτερα οχήματα τα υπάγουμε σε εθνικές αρμοδιότητες ή τα εξκαφικά κτλ. Μια σειρά από εξαιρέσεις με τις οποίες όμως δεν πάμε πουθενά τελικά. Και η δυνατότητα να ε, ορίσουμε συνθήκες πιο ε, αυστηρές ή να ξεπεράσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές ε, που ισχύουν στα κράτη-μέλη, υφίσταται. Μπορούμε να τις επαληθεύσουμε αυτό και έτσι να προχωρήσουμε. Χαίρομαι πάντως για αυτή την πρώτη συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές, πρώτη συζήτηση. Κάποια ζητήματα ε, επιμέρους έχουμε να τα διευκρινίσουμε ακόμα. Κυρία Σέναλοβα. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους οι οποίοι διευκρίνησαν τις τροπολογίες τους και σχολίασαν. Όπως είπε και ο κύριος Κούν, η θέση μας για τη νομική βάση που τελικά θα ζητήσουμε από το Συμβούλιο είναι κάτι πολύ βασικό. Ας επικεντρωθούμε τώρα στο περιεχόμενο των τροπολογιών και ας αφήσουμε το θέμα της νομικής βάσης για το δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Για τις τροπολογίες λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ συμφωνώ με αυτό το σύστημα διαβάθμισης κινδύνου που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν βλέπω γιατί να το φοβόμαστε. Αντίθετα, το είπα και στην αρχή. Και άλλοι συνάδελφοι το ανέφεραν. Το υποχρεωτικό ποσοστό είναι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε και το εύρος εφαρμογής, το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Σας ευχαριστώ και πάλι και προσβλέπω στη συνεργασία με τους σκιώδεις ηγητές επόμενες εβδομάδες. Παρακαλώ, κ. τρίτη συγγήτρια. Ευχαριστώ. με τον κύριο Μπράτμορν θα συνεχίσω τη συζήτηση, έφυγε βέβαια από εδώ, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι το άρθρο 1 δεν έρχεται σε αντίθεση με την ομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε αυξάνει το γραφειοκρατικό άχθος. Και αφού πρόκειται για οδηγία, πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια ρύθμιση για τη συμμόρφωση προς τα ε, κριτήρια. Δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες προβλέπουν ότι αν δεν έχει τον τεχνικό έλεγχο ένα αυτοκίνητο πρέπει να αποσύρεται. Εγώ δύο χρόνια έχω το αυτοκίνητό μου σε αυτή την κατάσταση και δεν ισχύει αυτό. Ούτε όλες οι χώρες σας ζητούν να φέρετε όλα τα έγγραφα μαζί σας στο τεχνικό έλεγχο. Τώρα στην κυρία Τικάου θέλω να πω ότι το άρθρο 1 σημείο 2 σίγμα ταφ υπάρχει. Κοιτάξτε το. Δεν νομίζω ότι έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ψηφίζουμε στις 30 Μαΐου. Επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων για τις οδικές ενδομεταφορές που περιλαμβάνει και την παρουσίαση δύο μελετών κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και ανάπτυξη και εφαρμογή των οδικών οδομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ να έρθουν εδώ οι προσκεκλημένοι. Κυρία Σάφισα, κλείστε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Thank you, Ms. We were all hearing your conversation. Όλοι ακούγαμε τι λέγατε εκεί στο πηγαδάκι γι' αυτό.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Η πρώτη παρουσίαση είναι της κυρίας Φρυσόνη που έχει να κάνει με την ανάπτυξη στην εφαρμογή του οδη... των οδικών εδωμεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, θα έχουν 15 λεπτά ο καθένας. Μην το πάρετε άσχημα, αλλά δεν έχω καταφέρει μέχρι τώρα κανένα να τον ε, πίσω να κρατηθεί μέσα στον χρόνο που του έχω δίνει. Το έχω δώσει. Λοιπόν, 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν την μελέτη αυτή για το, τις ενδομεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας παρουσιάσω το περιεχόμενο της έκθεσης που παρουσιάσαμε, τουλάχιστον το προσωρινό περιεχόμενο. Και εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στη δομή και θα ξεκινήσω με την εισαγωγή για να σας παρουσιάσω μετά τις αλλαγές που έχουν υπάρξει στον, στις ρυθμίσεις του τομέα αυτού και μετά θα περάσω στην εφαρμογή των κανόνων. Τέλος θα σας παρουσιάσω στοιχεία από τις έρευνες που έχουμε κάνει, χάρη βέβαια και στη συνεργασία που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στοιχεία που μας έδωσε. Τέλος, θα παρουσιάσω και τα αποτελέσματα υψηλού επίπεδου που ερευνήσαμε όσον αφορά τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης των μεταφορών αυτών. Ίσως να ξέρετε όλοι περί τίνος πρόκειται, πάντως σημαντικό είναι να επενθυμίσουμε ότι στην αγορά μεταφοράς εμπορευμάτων υπάρχουν βέβαια διαφορετικοί φορείς και τρόποι. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην μελέτη μας στις ενδομεταφορές. Στην, ε, στο σχέδιο αυτό βλέπετε ένας ε, Ιταλός που περνάει στη Γαλλία με τελική, τελικό προορισμό την Γαλλία. Ορίζεται η ενδομεταφορά σαν ε, κάποιον ο οποίος φεύγει από τη χώρα του και συνεχίζει σε μια άλλη χώρα μέλος. Υπάρχουν διαφορετικά είδη ε, μεταφορών εμπορευμάτων. Πέρα από τις εθνικές μεταφορές βέβαια που σίγουρα τις γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν ε, κεντρών ειδών διεθνεί. Και μία από αυτές είναι εδώ μεταφορές. Τους ορισμούς θα τους βρείτε στην παρουσίαση που νομίζω ότι σας έχει διανεμηθεί. Αυτό που είναι σημαντικό πάντως να δούμε πρώτα απ' όλα είναι ο ρόλος των μεταφορών επί του παρόντος στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι 1,2% σήμερα των υπηρεσιών μέσα στην Ευρώπη των 27 χωρών όσον αφορά τα εμπορεύματα. Υπάρχει διαφορά με τους 15 και τους 12. Στο μεταξύ των 12 έχει πιο δραστήριο ρόλο. Γενικά στις διεθνείς μεταφορές οι εθνικές μεταφορές είναι χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη το 12 από ό,τι στην Ευρώπη το 15. Και σε αυτό θα επανέλθω αργότερα όταν θα αναφερθώ στα δεδομένα που έχουμε από την αγορά. Να επενθυμίσω επίσης τις πιο σημαντικές αλλαγές στη ρύθμιση της αγοράς. Το 2009, όπως θα γνωρίζετε, πέρασε ένας νέος κανονισμός που διευκρίνιζε τους κανόνες που ρύθμιζαν την αγορά μέχρι τότε και κάλυπτε τα κενά και τις ελλείψεις και επιτρέπει σε μεταφορείς εμπορευμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετακινούνται σε άλλες χώρες βάσει μιας ε, προσωρινής, ε, προσωρινού διακανονισμού. Τα κριτήρια δεν ήταν όμως πολύ ξεκάθαρα ακόμα γιατί δεν υπήρχε ξεκάθαρος ορισμός για το τι σήμαινε temporary basis. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μετά από μερικά χρόνια συζητήσεων, πέρασε ένας νέος κανονισμός το 2009 που είχε στόχο να διευκρινίζει ακριβώς τους κανόνες και εισήγαγε πιο μετρήσιμα κριτήρια, ποσοτικά. Το περίφημο τρεις ε, δραστηριότητες σε 7 μέρες, που σημαίνει ότι μέχρι τρεις ενδομεταφορές θα μπορούσε να αναλάβει ένας μεταφορέας μέσα σε 7 ημέρες, από τη στιγμή που φορτώνει δηλαδή το φορτίο του. Ο κανονισμός αυτός επίσης φροντίζει και για μεγαλύτερη εναρμόνιση των απαιτούμενων εγγράφων, προκειμένου να αποδείξουν δηλαδή μεταφορές την ε, νόμιμη ενδομεταφορά. Θέλω επίσης να επιθυμίσω ότι ο κανονισμός αυτός πέρασε μέσα σε μια περίοδο που είχαμε μεγάλες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διεύρυνση πρώτα απ' όλα, 2004, κάτι το οποίο άλλαξε πάρα πολύ τις αγορές, άρα και τις εδώ μεταφορές. Υπήρχαν διμερείς περιορισμοί ανάμεσα στις παλιές χώρες μέλη και τις νέες χώρες μέλη. Πολλοί από τους περιορισμούς αυτούς βέβαια άρθηκαν το 2009. Και οι τελευταίοι περιορισμοί το 2012 που ήταν για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία νομίζω έπαψαν να ισχύουν. Αυτά σας τα λέω για να σας εξηγήσω ότι ο κανονισμός πέρασε σε μια περίοδο που είχαμε τεράστιες αλλαγές στην Ευρώπη. Τα βασικά ε, ζητήματα τα οποία εντοπίζονται με τον κανονισμό είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις όσον αφορά τους ορισμούς το multi-drops για παράδειγμα Άλλα προβλήματα έχουν να κάνουν με το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους ή και άλλα θέματα που είναι η ευθύνη των διαφόρων φορέων που δρούν αυτοί που για παράδειγμα φροντίζουν για την φόρτωση του φορτίου ή τα θέματα της ασφάλειας. Για να περάσουμε τώρα στο θέμα της εφαρμογής. Ο νέος κανονισμός βοήθησε την εφαρμογή των κανόνων, ακριβώς επειδή διευκρίνησε διάφορα πράγματα. Με την διευκρίνηση διευκρίνηση αυτή διευκρινίστηκαν και ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα πετούμενα έγγραφα και με τον έλεγχό τους από τις αρμόδιες αρχές. Παραμένουν όμως ζητήματα Για παράδειγμα, μερικές φορές είναι δύσκολο να ελέγξει κανείς τις παραβιάσεις. Για παράδειγμα, σε μια χώρα μέλος φορτώνεται ένα ε, φορτίο αυτό είναι δύσκολο να ελεγχθεί στη συνέχεια. Άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με τον συντονισμό ανάμεσα στις διάφορες αρχές υπεύθυνε με τον έλεγχο, είτε στην ίδια χώρα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. έχουν διαφορετικούς τρόπους για να εφαρμόζουν τους κανόνες οι χώρες μέλη και διαφορετική οργάνωση. Πολλές φορές υπάρχει και επικάλυψη στην ε, ευθύνη και στις αρμοδιότητες των αρχών των υπεύθυνων επιβάλλουν τον νόμο. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερο συντονισμός των δραστηριοτήτων των διαφόρων αρχών που επιβάλλουν τον νόμο. Έπειτα υπάρχει και το θέμα των ε, κυρώσεων. Και αυτό μας δυσκολεύει. Οι παλιές χώρες μέλη είναι εκείνες, χώρες μέλη είναι εκείνες οι οποίες αναλαμβάνουν να επιβάλλουν και τις κυρώσεις. Η χώρα στην οποία κυκλοφορεί δηλαδή το φορτηγό. Καλύτερη εναρμόνιση της εφαρμογής είναι κάτι που χρειάζεται εξαιτία του μεγέθους που διαφέρει στις αρχές που επιβάλλουν τον νόμο. Τέτοια πράγματα σημαίνουν ότι η πιθανότητα, ο κίνδυνος δηλαδή να πιαστεί κάποιος που παραβαίνει τους κανόνες διαφέρει από χώρα σε χώρα επειδή ακριβώς η εφαρμογή του, της ρύθμισης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σας είπα θα επανέλθω στην αγορά. Στην αγορά λοιπόν υπήρξε αύξηση των δραστηριοτήτων μεταφορέ εμπορευμάτων ενδο, μεταφορές δηλαδή από 14 σε 19 εκατομμύρια τόνους το χιλιόμετρο ανάμεσα στο 2006 και το 2011. Όπως επίσης υπάρχουν και διαφορές στα εμπορεύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 12, πέρασε από 12% το 2006 στο 40% το 2011. Με την ε, η Πολωνία σε ηγετική θέση. Ίσως γιατί έχουν αρθεί οι περιορισμοί που υπήρχαν παλιότερα στην Ευρώπη των 12 και των 15. Αναλύοντας πάντως τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, διαπιστώνουμε ότι το βασικό σε αυτά που ερευνήσαμε είναι η διεύρυνση. Η διεύρυνση ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η μεγάλη αλλαγή και η άρση των φραγμών και των εμποδίων. Είναι βέβαια κάτι που είχε θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Μεταξύ των 15, το θετικό είναι ότι έχει μειωθεί το κόστος. Οι χαμηλές τιμές ωφελούσαν τη βιομηχανία στην Ευρώπη των 12. Τώρα αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι έχει μειωθεί το κέρδος. ή οδηγεί. πολλές φορές είναι αυτό ασχολούμε και όχι μόνο βέβαια στην περίπτωση των ενδομεταφορών. Στο μέλλον δηλαδή μπορεί να υπάρξουν κάποιες ελλείψεις. Έπειτα, ασφάλεια. Και αυτή βέβαια απορρέει από τις αλλαγές που έγιναν. Συνολικά πάντως είναι σαφές ότι οι ανισορροπίες που υπάρχουν στην κοινωνική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη και ο διαφορετικός τρόπος εφαρμογής και των εδώ μεταφορών και όχι μόνο, είναι μία πρόκληση για τον ανταγωνισμό. Η πρόκληση αυτή είναι εκείνη που μας οδηγεί και στα συμπεράσματά μας. Εδώ στα συμπεράσματα προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις. Σκεφτήκαμε ότι πρώτα απ' όλα έπρεπε να εντοπίσουμε τους κύριους στόχους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο βασικός στόχος είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή η μείωση των ταξιδιών χωρίς φορτίου και η δημιουργία ενός ε, ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών. Αυτοί οι δύο στόχοι βέβαια πρέπει να μετρηθούν, μάλλον πρέπει να πραγματοποιηθούν με διαφορετικά μέτρα, με μελέτες αντικτύπου και επειδή βέβαια μου έχετε βάλει και περιορισμό στο χρόνο, θα σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το στόχο της αποτελεσματικότητας. Εμείς προτείνουμε διαφορετική προσέγγιση από τη σημερινή. Για το θέμα των, ε, του ανώτατου αριθμού ε, διαδρομών, το 3 που είχαμε. Ίσως τους κανόνες θα έπρεπε να τους εφαρμόζουμε με τέτοιο τρόπο που να λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη μας τις διαδρομές που κάνει το έχουμε και όχι περισσότερο το πόσες φορές φορτώνεται. Η χρήση επίσης του GPS και άλλου εξοπλισμού είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της διαδρομής των φορτηγών, πότε περνά τα σύνορα δηλαδή. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, μήπως υπάρχουν τέτοια συστήματα που μπορούν να εγκατασταθούν. Και όσο για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφοράς, η σύστασή μας είναι ότι αν ανοίξει περισσότερο το σύστημα χρειάζεται και μεγαλύτερη εναρμόνιση, ιδιαίτερα στον τομέα των πρακτικών, των ε, προδιαγραφιών όσον αφορά την εργασία, και η προσέγγιση που εμείς συστήνουμε ευθυγραμμίζεται σε αυτήν που πρότεινε το 2002 η ομάδα υψηλού επίπεδου. Δηλαδή να είναι σταδιακή και ελαστική. Το άνοιγμα της αγοράς δηλαδή να γίνεται σταδιακά και με ελαστικότητα. Ευχαριστώ. πολύ έξι δεύτερα παραπάνω, αλλά εντάξει θα το δέχομαι. Κύριε Παστόρη, παρακαλώ να μας κάνετε τη δική σας παρουσίαση. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Θα μιλήσω Ιταλικά. Δράτω με τις εξαιρετικές ευκαιρίες ε, που έχουμε για υπηρεσίες διερμηνίας, οπότε θα μιλήσω στην Ιταλική γλώσσα. Λοιπόν, η δεύτερη μελέτη θα σας παρουσιάσω αφορά κατά κύριο λόγο τις ε, συνθήκες εργασίας και τις ε, κοινωνικές ε, συνθήκες που διέπουν τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων και συνδέεται δηλαδή τροποντινά με το θέμα των οδικών μεταφορών και θα δούμε με ποιο τρόπο. Λοιπόν, στην παρουσίαση που θα κάνω, προσπαθώντας να θεωρήσω το χρόνο των 15 λεπτών, όπως η συνάδελφος, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε κάποιες ενδείξεις από ποιο το σημείο εκκίνησης για αυτή τη μελέτη και μετά θα δούμε τις δραστηριότητες που κάναμε στα πλαίσια της μελέτης, που ήταν ουσιαστικά να ορίσουμε ποια είναι, ποιο είναι το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που θα εξετάσουμε, με, ποιες, ε, με ποια αποτελέσματα που έχει δώσει ως σήμερα. επειδή θα αξιολογήσουμε τις συνθήκες ε, εργασίας και τις ε, κοινωνικές συνθήκες με οποίες εργάζονται οι οδηγοί και τα κρίσιμα ζητήματα σε ό,τι αφορά την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών και το θέμα του καποτάζ των ενδομεταφορών δηλαδή που είναι και το βασικό θέμα αυτής της ακρόασης. Λοιπόν, αν η στόχη αυτής της μελέτης είναι εξή. Ε, να δούμε τροποντινά και γενικότερα τις συνθήκες εργασίας των οδικών και τα επίπεδα ελέγχου που διενεργούνται σήμερα στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Να αναλύσουμε την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία μεταφράζεται στις εθνικές νομοθεσίες και να δούμε και το θέμα της εφαρμογής ως ιδιαίτερο στοιχείο που συνδέεται και μια προηγούμενη μελέτη που είχαμε εκπονήσει και αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και να αναφέραμε στον κανονισμό, εφαρμογή του κανονισμού 561 του 2006 και τα κρίσιμα στοιχεία που συνδέονται με τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών βαρέων οχημάτων. Μεθοδολογικά εστιάσαμε τη μελέτη και σε άμεσα στοιχεία, πέρα δηλαδή του βιβλιογραφία και την ίδια την νομοθεσία, προσπαθήσαμε να δούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να ακούσουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους stakeholders. Κάποιοι εξ αυτών είναι παρόντες και εδώ σε αυτή την αίθουσα αλλά και άμεσα τους ίδιους τους επαγγελματίες οδηγούς για να ακούσουμε από πρώτο χέρι την άποψη αυτόν τον ανθρώπων, δηλαδή πώς εισπράτεται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους ε, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εδώ βλέπετε την απαρίθμηση των νομοθετικών πράξεων που λάβαμε υπόψη στη μελέτη μας, ιδίως τις οδηγίες που αφορούν τους χρόνους οδήγησης και χρόνους ανάπαυσης, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η νομοθεσία. Είναι και, η άλλη οδηγία για το χρόνο εργασίας γενικότερα, όπως και τους κανόνες των κανονισμών 1071 και 1072 του 2009. Όταν μιλάμε για συνθήκες εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη και πολλές άλλες οδηγίες που δεν εκπονήθηκαν συγκεκριμένα για να ρυθμίσουν αυτό το κλάδο, αλλά συνδέονται και περιέχουν σημαντικές διατάξεις που αφορούν και αυτούς τους εργαζόμενους, όπως είναι οι αποσπασμένοι ή εποχικοί εργαζόμενοι. Αν δούμε τώρα πιο γενικά το θέμα που κάνουμε μια επισκόπηση, θα δούμε ότι το ευρωπαϊκό τοπίο άλλαξε σημαντικά καθώς και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και περισσότερο άνοιγμα στον ανταγωνισμό ανάμεσα στους επόρους. Αν δούμε όμως κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα, θα δούμε ότι οι συνέπειες ήταν και κάποιες περιπτώσεις αναπάντεχες. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια έχουμε τη σύνοψη όλων των νομοθετικών πράξεων που λάβαμε υπόψη με πορτογαλίνι οδηγίες, με γαλάζιο ή κανονισμοί. Σε ό,τι αφορά την ε, νομοθεσία, το είπα και πριν, ακολουθήσαμε δύο οδούς ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη βελτίωση των κοινωνικών προτύπων ε, για τους εργαζόμενους, ό,τι αφορά το χρόνο εργασίας, χρόνους οδήγησης, χρόνους ανάπαυσης κτλ. Αλλά και ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, ο άλλος στόχος ήταν η δημιουργία, η πραγωγή ενός ε, πεδίου ίσου ανταγωνισμού και θεμητού ανταγωνισμού στον τομέα των ε, οδικών μεταφορών. εντοπίσαμε ως πολύ ισχυρό στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό τον κλάδο εργασίας στην Ευρώπη και το ανέφερε και οι συνάδελφους, είναι το μερίδιο της αγοράς ε, των επαγγελματιών ε, της Ευρώπης των 12, δηλαδή των νέων κρατών μελών, που προσχώρησαν στην Ένωση με το 2004 οδήγησε στην ε, εισρωή ενός πολύ σημαντικού αριθμού επαγγελματιών ε, του κλάδου. Αυτό δεν σημαίνει και εναρμόνιση ε, της αγοράς σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών. Αντίθετα βλέπουμε σημαντικές διαφορές, μεγάλες διαφορές και έτσι βαθύνθηκε το χάσμα ανάμεσα στην κατάσταση που βλέπαμε πριν στην Ευρώπη των 15 σε σχέση με το τι βλέπουμε στην αγορά της Ευρώπης των 12. Βλέπουμε και μακροοικονομικές σημαντικές διαφορές, δηλαδή σε επίπεδο αμοιβών, αλλά και σε επίπεδο γενικότερο εργασιακού πλαισίου, όπως ισχύει σε κάθε χώρα. Αυτές οι διαφορές και οι ανισότητες οδήγησαν σε προσπάθεια εξέβρεση λύσεων και από τους ίδιους ε, τους εμπόρους, ε, τους επιχειρηματίες μεταφορές, για να μπορούσαν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά. Ε, μια προσπάθεια επιβολής ρυθμίσεων, ώστε να μπορεί να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, Άρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ισότητα και πιο προσπελάσιμη αγορά για όλους, αλλά ταυτόχρονα υπήρξαν και άλλες συνέπειες, αρνητικές συνέπειες, αναφέρθηκαν ε, ήδη κάποιες αρνητικές συνέπειες, θα πούμε και σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες όπως είναι η εταιρεία Letterbox, ε, η, η ψευδή δήλωση ε, μισθωτών εργαζομένων ουσιαστικά ως αυτοαπασχολούμενοι ή οι ψευδείς δηλώσεις ό,τι αφορά το ωράριο εργασίας. Η χρήση αφορα τωρα εργασια αυτών των ε, αθέμητων πρακτικών με στόχο να γίνει κανείς πιο ανταγωνιστικός μειώνοντας το κόστος ε, μεταφοράς ώστε να ανταποκριθεί κανείς ε, και στις ανάγκες ε, του πελάτη οδήγησαν στην επιδίνωση των συνθήκων εργασίας και διαβίωσης των επαγγελματιών οδηγών. Δεν ανταποκρίνεται γρήγορα το μηχάνημα. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο μιλητή. Σε ό,τι αφορά τις συνδίκες εργασίας, ε, ανέφερε και πριν ότι υπάρχουν ανισότητες. Στην Ευρώπη των 12 τα επίπεδα των μισθών κατά μέσο όρο ε, είναι χαμηλότερο από την Ευρώπη των 15. Κατά μέσο όρο, παραλαμβάνω, μην γενικεύουμε υπερβολικά. Σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα, το προφίλ εργασίας, ζητείται όλο και περισσότερη ευελιξία στην εργασία και παροχή υπηρεσιών που δεν είναι καθαρά η οδήγηση, αλλά και άλλες υπηρεσίες, όπως ε, η παρακολούθηση της φόρτωσης εκφόρτωσης, όπως επίσης είναι και χρόνοι αναμονής, που προσμετρούνται στο χρόνο ανάπαυσης. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των στοιχείων οδηγεί σε μια γενικότερη μείωση ε, των επιπέδων ε, των αμοιβών. Να δούμε τώρα ποια είναι τα στοιχεία τα, στα οποία καταλήξαμε άμεσα από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους οδηγούς Δυστυχώ δεν μπορώ να σα δείξω, δεν προλαβαίνω να σα δείξω όλε τις διαφάνειες, αλλά τα κύρια στοιχεία θα σας δείξω εδώ που αφορούν κύρια στοιχεία, όπω είπα, που επηρεάζουν τι συνθήκε εργασία και διαβίωση των επαγγελματιών οδηγών. Βλέπουμε ότι είναι συνθήκε απασχόλησης, το ωράριο, το ίδιο το ωράριο εργασίας, Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που υποδεικνύουν οι ίδιοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ως στοιχεία κλειδιά. Μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που θεωρούν θεωρούν οι ενδιαφερόμενοι ότι έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια είναι αυτά που συνδέονται με το εργασία, όπω είπα και πριν, με τα επίπεδα ε, των αμοιβών και με τι συνθήκες εργασία. Γιατί βλέπει κανεί ότι ε, ζει σε, και εργάζεται σε ένα όλο και πιο επισφαλές περιβάλλον. Άλλα στοιχεία κλειδιά στα οποία καταλήξαμε, έτσι για να πάρετε μια ιδέα, μια μετρήσιμη αν θέλετε ιδέα, ε, κάποια ποσοτικά στοιχεία του αντικτύπου. Στην Ευρώπη των 12 βλέπουμε ότι ο μέσος μισθός ε, κυμαίνεται ανάμεσα στα 250 με 450 ευρώ το μήνα. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλα επιδόματα μεταφορά 40 με 45 ευρώ την ημέρα, αλλά ε, ε, ο επαγγελματίας οδηγός θα πρέπει να ζει σε μια επισφαλή κατάσταση ουσιαστικά. Γιατί ουσιαστικά ζει μέσα στο ίδιο το φορτηγό όχημα, εκεί ε, τρώει, ο οδηγός εκεί κοιμάται όλο και διευρύνονται ε, τα, ε, η εφαρμογή των συστημάτων πληρωμής αναπαραχή, δηλαδή ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύει ο οδηγός, ένα σύστημα δηλαδή που κανονικά δεν προβλέπεται στις ε, συμβάσεις έργου, Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και επιπρόσθετες σε ό,τι αφορά την ιατρική περίθαλψη, και λοιπές παροχές. Γενικότερα δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρότερα προβλήματα και αντιμετωπίζουν και διεκριτική μεταχείριση λόγω εθνικότητας κάποιες φορές ε, και βλέπουμε ε, κάποια δικαιώματά τους ό,τι αφορά ε, επιδόματα άδειες και διακοπών δεν τηρούνται πάντοτε συνθήκες ασφάλειας ε, στους χώρους ε, στάθμευσης, εκεί δηλαδή που μετά το τέλος του χρόνου εργασίας ε, σταματούν και σταθμεύουν οι οδηγοί. Πρέπει να είναι και προσεκτικοί να μην υπάρξει κάποια κλοπή, γιατί είναι υπεύθυνοι για το φορτίο που φέρουν. Είναι υπεύθυνοι και για το όχημα, για το καύσιμο και για το φορτίο που φέρουν. Τώρα, ποια είναι τα πλέον κρίσιμα στοιχεία. Ε, γιατί, ναι, μεν υπάρχει νομοθεσία, κάποιες πρακτικές ε, έχουν κατακριθεί, κάποιες ε, πρακτικές επίσης θεωρούνται ότι είναι στα όρια, είναι στο borderland και εκεί είναι το, το πρόβλημα, τι είναι παραδεκτό, ε, ή τι όχι, τι είναι, αλλά κατά πόσο η τι οχι τι αλλα κατα ποσο είναι πρακτικη letterbox ή ε, οι πρακτικές flagging out είναι αποδεκτές ή όχι. Επίσης η μεταφορά των υπηρεσιών σε τεχνη... σε εταιρείες βιτρίνα που έχουν την έδρα τους ε, σε χώρες με πολύ πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ δύσκολο. Και αυτό αφορά και τον ίδιο τον έλεγχο, καθώς αυτό το στοιχείο κλειδί είναι ότι χρησιμοποιούνται οδηγοί από τις χώρες των 12 στις χώρες των 15, όπου απασχολούνται και για μακρές περιόδους, χωρίς δηλαδή να τηρούν τις υποχρεώσεις ε, που, ε, που προβλέπει η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Δηλαδή, δεν προσαρμόζουν τις συνθήκες εργασίας και τον ώρα εργασίας στις χώρες στις οποίες παρέχεται υπηρεσία, με άλλα λόγια. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, το καποτάζ έχουν ακουστεί ήδη διάφορα. Έχουμε να κάνουμε μια, τις πιο μεγάλες αγορές όπου υιοθετούνται πρακτικές αποδεκτές σε ένα βαθμό. Επειδή όμως οι μεταφορές, οι οδικές μεταφορές είναι πολύ μεγάλη αγορά, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι έχουμε ενδελεχείς ελέγχους ε, και αυτό το φάνηκε και στην προηγούμενη μελέτη. Για να πάρετε μια εικόνα με αριθμητικά στοιχεία στην Ιταλική περίπτωση. Μείωση του κόστους κατά 20-25% χρησιμοποιώντας υπαλλήλου από αυτές τις εταιρείες Letterbox, όπως και εταιρείε συνδυασμένων μεταφορών που δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν ξέρω αν έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Το ξεπέρασα? Σε 15 λεπτά? Όχι, όχι, το ξεπεράσατε, λέει ο πρόεδρος. Ε, φτάσα στα συμπεράσματα. Για να κλείσω, λοιπόν, θέλω να πω ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει στην ε, ευρωπαϊκή αγορά οδικών μεταφορών ανάγκασαν ή κάλεσαν ε, και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να παρακολουθήσει αυτές τις αλλαγές ώστε να προφυλαχθούν κάποια πρότυπα ε, στην συνθήκη εργασία, αλλά και ταυτόχρονα να διαφυλαχθεί και ο ανταγωνισμός. Παρά αυτά, υπάρχουν πολλές διαφορές και είμαστε πολύ μακριά από το να πούμε εναρμόνιση των συνθηκών εργασίας, δηλαδή το λόγιων συνθήκες εργασίας μιλώ για συμβάσεις εργασίας και τους όρους ε, των συμβάσεων αυτών. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής ε, Κοινωνικής Νομοθεσίας, καταγράφουμε μία έλλειψη κοινή ερμηνεία ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις πρακτικές και τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Εδώ όμως θέλω να επιμείνω και να πω ότι η εφαρμογή νομοθεσία συνεπάγεται και ε, ένα οικονομικό κόστος για τα κράτη-μέλη. Δεν είναι εύκολο να μιλάμε για εφαρμογή νομοθεσία. Συνεπάγεται κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μεταξύ των συστάσεων, αυτά αρκετά, λέει ο πρόεδρος. Αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια, λέει ο μιλητής. Συστάσεις πρέπει να βελτιωθεί στην εργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχει έλεγχος ε, της συμπεριφοράς σε όλα τα κράτη-μέλη, άρα εναρμόνιση εν προκειμένου του ελέγχου, δημιουργεί ίσως ενός μητρώου των εταιριών που δεν τηρούν τους κανόνες, ε, ένα, ενός κοινού συστήματος ε, ε καταγραφής του κινδύνου, και βελτίωση των πρακτικών εφαρμογής της νομοθεσίας κατά παρόμοιο τρόπο με αυτό που έγινε για την οδηγία 22 του 2006 που αφορά τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης. Ελπίζω όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης να τα βρείτε στην μελέτη που σας διανύμαμε και είμαι στη διάθεσή σας για πιθανές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Can τη χάρη να κλείσετε το μικρόφωνο σας. Αγαπητοί φίλοι, ο χρόνος μας τρέχει. Έχουμε τώρα ερωτήσεις και απαντήσεις. Ε, και επισημαίνω ερωτήσεις και απαντήσεις, όχι ερωτήσεις μεταλογιδρίου, στις οποίες ε, δίνονται απαντήσεις μεταλογιδρίου. Παρακαλώ λοιπόν, ερωτήσεις σύντομα και ουσιαστικά για να γίνει και η ανταλλαγή απόψε με τους κοινωνικούς εταίρους. Ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει πρόβλημα όταν έρχεται κανεί να παρουσιάσει την έκθεσή του. Εσεί, κυρία Φριζόνη, αποτελείτε λαμπρή εξαίρεση. Ο κύριο Κούν έχει τον λόγο. Ναι, πρόεδρε. Και εγώ πολύ σύντομα. Η διεύρυνση αυτών των ενδομεταφορών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω είναι κάτι το ενδιαφέρον, δεν υπάρχει λόγος να, να μη συμφωνήσουμε. Για τον κύριο Παστόρη, θα ήθελα να ρωτήσω εάν όντω στις οδικές μεταφορές των κρατών μελών υπάρχουν προσλήψεις εργαζομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έρχονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους να δουλέψουν μέσα στη βδομάδα, δεν έχουν μερικές φορές καν στέγη, ε, δουλεύουν μόνο μέσα στο φορτηγό, δεν έχουν χρόνους ανάπαυσης, ε, να από τη μια διαδρομή στην άλλη και δεν τηρούνται οι κοινωνικές ε, συνθήκες τις οποίες έχουμε ήδη απαιτήσει και εξασφαλίσει για την εσωτερική αγορά. Όταν υπάρχουν συνθήκες επασχόλησης, όταν υπήρχε συνθήκη Σέγγεν, είναι αδύνατον εμείς να δεχθούμε περαιτέρω άνοιγμα στην ε, ενδομεταφορά, στις ενδομεταφορές, στο καμποτάζ, εάν προηγουμένως δεν έχουν υλοποιηθεί οι ε, νόμοι που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν υπάρξει εναρμόνιση τη εθνική νομοθεσία. Ευχαριστώ κύριος Αλκαντράου. Παρακαλώ ερωτήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις, για τις μελέτες, χρήσιμες για τη συζήτηση και τα συμπεράσματά σας είναι σαφή. Ελευθέρωση, αλλά συγχρόνως κοινωνική εναρμόνιση. Οι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Τα τελευταία χρόνια ξέρουμε τι έχει συμβεί με τις αποσπάσεις, Η καταχώρηση επιχειρήσεων που πρέπει να είναι προσβάσιμες σε επιθεωρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι σε κατάλογο ανοιχτό. Για τον ταχογράφο επίσης έχουμε συζητήσει πολύ και εμεί θέλουμε να βελτιωθούν οι έλεγχοι. Έχω πάντως μια ερώτηση προς τους δυο σας. Λέτε ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα για την κοινωνική εναρμόνιση. Ας υποθέσουμε ότι εσείς πρέπει να φτιάξετε την νομοθεσία. Τι θα βάζατε σαν δύο προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τους εργαζομένους και συγκεκριμένα βέβαια έτσι για να μπορέσουμε να εμπνευστούμε από αυτά που θα μας πείτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους δύο αγορητές για την καλή δουλειά. Για τη δική μας καλή δουλειά καλό είναι να έχουμε τη δυνατότητα της ε, αναφορά σε τέτοιου μελέτε μελέτες και ότι φοβούμε ότι αυτό μπορεί να εξυπηρετεί μόνο το στόχο της ε, αρχιοθέτηση. να γεμίσουμε ράφια, γιατί πολλές τέτοιε μελέτες υπάρχουν. Συγκεκριμένες ερωτήσεις, αντίστοιχε με αυτές του κ. Αλχαντράουη. Πριν από κάποια χρόνια στην έκθεση Ράνερ είχαμε μιλήσει για διαφορετικούς ελέγχους, για ελλειπείς ελέγχους για απουσία κυρώσεων, για προβλήματα ως προς την υπερσυνοριακή επιβολή κυρώσεων ή ποινική δίωξη και μας είπε ο κύριος Κάλλα σήμερα το πρωί ότι κάποιοι από τους νέους ελέγχους δεν μπορούν να αξιολογηθούν θελητικά. Αμφιβάλλω εγώ, αλλά μπορείτε όντως να αξιοποιήσετε αυτό το νομοθέτημα, γιατί έχει αλλάξει το μεταξύ νομική βάση, για μια καλύτερη αστυνομική συνεργασία. Μπορείτε να στηριχθείτε σε αυτή την αστυνομική συνεργασία για να βελτιωθεί ο έλεγχος πέρα από το τομέα του καποτάζ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριος Μπισέπ. Και ευχαριστώ πολύ για τις ε, εκθέσεις που παρουσιάσατε. Όταν λέτε ότι πρέπει να ανοίξει παραπάνω το σύστημα των μεταφορών, δικό των μεταφορών και οι έλεγχοι να ενισχυθούν, νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι ποτέ, ακόμη και αν ε, πολλαπλασιάσουμε, πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των ε, υπαλλήλων που θα υποφορτιστούν με τον ε, έλεγχο αυτών, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε ουσιαστικούς ελέγχους όταν τομέα του αριθμού των ε, φορτηγών οχημάτων που βρίσκονται στους δρόμους μας. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, ε, δεν συμφωνείτε ότι όσο δεν υπάρχει ένα αρμονισμένο κοινωνικό πλαίσιο στην Ευρώπη, το οποίο θα προσδιορίζει συνθήκες πολύ σημαντικές που αναφέρατε και εσείς, όπως ελάχιστο μισθό, που να ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινωνικούς κανόνες και συνθήκες ε, χρήσης για ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν αυτές ε, οι δυνατότητες για έλεγχο, δεν πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει να ανοίξει περισσότερο το καποτάζ. Αντί γι' αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τις, ε, τα μέσα σταθερής τροχιάς και όχι να ρίχνουμε περισσότερα φορτηγά πάνω στους δρόμους μας. Ευχαριστώ κύριο Ρικέ και ευχαριστώ πολύ τους δύο συγγητές που μας μίλησαν ξεκάθαρα για, τον, για το σχετικά περιορισμένο πλέον έκτημα από, το, από την απελευθέρωση του με τίμημα αίμα και δάκρυα προς, τις κοινωνικές, προς την κοινωνική προστασία, στο κοινωνικό επίπεδο δηλαδή, χιλιάδες οδηγών φορτηγών που έχασαν τη δουλειά τους και αντίστοιχα χιλιάδων σκλάβων που είναι πάνω στους δρόμους και που δουλεύουν σε όρους απαράδεκτος κατόπιν, κατόπιν ε, της θέσπισης ευρωπαϊκού νομοθετήματος. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι μια από τις πιο ε, πύριες νίκες που έχουμε εξασφαλίσει με μια ε, οδηγία Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο, εάν έρθει αυτή η πρόταση για το καβατάζ, θα επιοφεληθεί για να την καταργήσει, να καταργήσει το άνοιγμα. Έχω μια ερώτηση, χιλιάδες τα είχα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε με κάτι. Θεωρείτε ότι μπορούμε με τρόπο αυστηρό και τυπικό να εφαρμόσουμε το καθεστώς του αποσπασμένου εργαζομένου σε όλους τους μεταφορείς που εργάζονται και κάνουν τις ενδομεταφορές ε, και με αυτό βέβαια δεν λύνεται το πρόβλημα των ελέγχων. Ευχαριστώ, Τιτσό. Σύντομα, Σίλβια. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και από τις ε, μελέτες που παρουσιάστηκαν αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το κύριο πρόβλημα των οδηγών είναι ο χρόνος ε, οδήγησης, ο χρόνος ανάβαυσης και η τήρησή τους. Στον ψηφιακό ταχογράφο είχαμε προσπαθήσει ε, με την ευκαιρία της συζήτηση να καλέσουμε στην επιβολή κυρώσεων, με αντίσταση όμως μεγάλη από τα κράτη-μέλη και πρέπει να επανέλθουμε. Πώς μπορούν όμως να εναρμονιστούν οι κυρώσεις, για τα κράτη-μέλη αντιτίθενται και ρωτώ πόσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί κυρώσεις. Εσείς επισημάνατε αρκετά προβλήματα, αλλά από την πλευρά του ελέγχου πόσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί κυρώσεις. Ήταν αρκετά σοβαρές αυτές οι κυρώσεις για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Ασφαλέστερα, ε, ασφαλέστερα χώροι στάθμευση παραδείγματι υπάρχουν γιατί αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό λόγο να μην τηρηθούν οι χρόνοι οδήγηση ανάπαυση από τον οδηγό. Επίση στην, στην Γερμανία υπάρχουν εταιρείε οι οποίε χρησιμοποιούν οδηγού από τι Φιλιππίνες για έξι μήνε και για τις διεθνείς οδικές μεταφορές, υπερεθνικές καλύτερα μεταξύ των κρατών μελών. Και άρα έχουμε χώρες οι οποίες ενθαρρύνουν ή ευνοούν την απασχόληση εργαζομένων μη διαμενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαμηλού κόστους, low cost, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η Γερμανία δεν γνώριζε καν τον ελάχιστο μισθό. Ως εκ τούτου κάποια στοιχεία νομίζω πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω. Εγώ είμαι υπέρ της απελευθερώσης των ενδομεταφορών, είμαι υπέρ της κατάργησης των φραγμών στις ενδομεταφορές, διότι η απελευθέρωση αυτών, κατά την άποψή μου, θα φέρει σταδιακά καλύτερες ε, συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικής, ε, κοινωνικές συνθήκες. Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λίχτενμπέργκερ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συστήσει πολύ για την επιβολή των κανόνων και κυρίως των χρόνων άπαυσης και οδήγησης. Και δεύτερον, και ερωτώ λοιπόν τι έχει γίνει με αυτό και δεύτερον έχει μελετήσει ε, ο ένας ή ο άλλος ομιλητής τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί και πόσο αποτελεσματική ήταν η διεξαγωγή των ελέγχων αυτών ως προς την παρακολούθηση των ενδεχομένων αδικημάτων που διαπιστώθηκαν. διότι διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν πουθενά ένοχοι για τίποτα, αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώ. Δεύτερον, ε, το καμποτάζ, αν δεν μεταφορέ, ε, υποστηρίζονται από κάποιου με το επιχείρημα ότι αποφεύγουμε την κυκλοφορία των ε, φορτηγών με άδειο φορτίο. και μετά μα λέτε ότι δεν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχει έλεγχο, δεν υπάρχει. Το εχογράφο ελέγχεται νέου. Ναι και αν ελέγχεται, θέλουμε τα στοιχεία. Εάν όμως δεν υπάρξει περιορισμός του, ε, της κυκλοφορίας φορτηγού ε, χωρίς φορτίο, του άδειου φορτηγού δηλαδή, τότε γιατί θα πρέπει καθημερινά να υποβαθμίζονται τα δικαιώματα τα εργασιακά των ε, εργαζομένων στον τομέα αυτών χωρίς κανένα πλέον έκτημα. Είναι πολύ σαθρή αυτή η λογική. Ευχαριστώ στο Γόρμα. Από Σύρο την, ε, το έτοιμο, Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάνσινας. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακολούθησα και διερωτώ με αν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρούμε λύση για την απελευθέρωση του ίσεν των δεματοφορών γιατί φαινόμενο μπορεί να είναι εύστοχη λογική λύση, η εσωτερική αγορά σημαίνει και ε, ε μεταφορές σε όλη την Ευρώπη χωρίς εμπόδια, αλλά ε, διερωτώμεθα αν θα τα καταφέρουμε. Όταν οι κοινωνικέ συνθήκε στα κράτη-μέλη είναι τόσο διαφορετικέ από τη μία περιφέρεια, μάλιστα στην άλλη, μέσα στο ίδιο κράτο μέλο. Και διερωτώμε αν θα τα καταφέρουμε. Οι πολλέ συστάσει που μα διατυπώσατε, πιστεύετε ότι μπορούν να υλοποιηθούν. Εσεί ίδια πιστεύετε ότι μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από μια νομοθετική διαδικασία και με συμφωνία των κρατών μελών. Βλέπετε κάποια ευκαιρία, πιθανότητα να γίνει αυτό και εάν ναι, πότε. Ευχαριστώ και μια ερώτηση από μένα, λέει ο κύριος Σίμψον. Θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε, παρακαλώ, όσον αφορά τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αυτών που μεταφέρουν ε, εμπορεύματα στην Ευρώπη. Δεν είναι ίδιες βέβαια όπως είναι στη Λατινική Αμερική που έχουν τη σάνδηση στην Αφρική γιατί αυτά που διαβάζω εγώ εδώ μου θυμίζουν περισσότερο ότι είναι ποσαχάρη Αφρική με κάθε σεβασμό που έχω σε αυτούς και έχουν να κάνουν με που προσπαθούν να περάσουν τις άνδε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαντάζομαι ότι είναι διαφορετική κατάσταση. Ίσως ε, θα έπρεπε την Διεθνή Οργάνωση Μεταφορέων να ρωτήσουμε. Εσείς κύριε Φριζόν έχετε και να μας πείτε, κύριε Φριζόν να μας απαντήσετε. Ναι για τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες περισσότερο θα έπρεπε να απαντήσει ο συνάδελφος. Εγώ θα αρχίσω από την τελευταία ερώτηση. Κάνουμε συστάσεις που έχουν να κάνουν με τους στόχους αποτελεσματικότητας, για παράδειγμα. Γιατί, ναι, πιστεύω ότι μπορούν να εφαρμοστούν αυτοί οι στόχοι. ο αριθμός των ε, τριών ε, δράσεων σε μία εβδομάδα. Ναι, κάποια πράγματα που μπορούμε να χειριστούμε. Αυτές είναι οι συστάσεις μας. Τώρα, για το γεγονό ότι υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι αλήθεια. Η ελευθέρωση και όχι μόνο, γενικά η διεύρυνση μας οδηγεί για παράδειγμα σταδιακά σε ίδια επίπεδα μισθών. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχουν διαφορές στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, κάτι το οποίο φάζει και το θέμα της εφαρμογής της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Στη μελέτη μας το αγγίζουμε και αυτό είδαμε ότι η οδηγία αυτή εφαρμόζεται πολύ δύσκολα στις εδωμεταφορές. Ορισμένες χώρες προσπαθούν, όπως η Γαλλία. Το κατά πόσο εφαρμόζεται με το σωστό τρόπο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Φαίνεται ότι είναι δύσκολη η σωστή εφαρμογή. Οι συστάσεις μας λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι το οποίο να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει και όχι απλώς να λέμε εντάξει θα το εφαρμόζουμε και ας μην λειτουργεί. Το θέμα τώρα της καταχώρησης των επιχειρήσεων, δεν θυμάμαι ποιος το ρώτησε. Θέλουμε βελτίωση της κυκλοφορίας των πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι εδώ είναι ένα παράδειγμα όπου κάποια καταχώρηση χρειάζεται ξένων επιχειρήσεων και έχει να κάνει πάλι και με την οδηγία για τους αποσπασμένους. Στη δικιά μας την ανάλυση πάντως φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες. Και πάλι χρειάζονται πρακτικές λύσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο. Με πάση περιπτώσει, ό,τι ερωτήσεις έχετε, ευχαρίστω θα σας απαντήσουμε. Ε, Ο κύριος Παστόρε. πολλά, πολύ εύστοχα όλα τα ερωτήματα. Εδώ δεν θέλουμε να σας δείξουμε ή να σας αποδείξουμε ότι έχουμε μια αγορά οδικών μεταφορών κακής ποιότητας. Απλά είναι πολύ γρήγορη η μετάβαση και ε, παρά τα αυτά είμαστε πολύ μακριά ακόμη από την εναρμόνιση. Αυτό προσπαθούσα να πω. Δηλαδή με το άνοιγμα που έγινε ε, στα νέα κράτη-μέλη βιώσαμε μία ταχύτατη μετάβαση στις σημερινές συνθήκες ε, εργασίας. Και μια ταχεία μετάβαση και ταχεία επιδείνωση των συνθήκων μια ραγδαία επιδείνωση των συνθήκων εργασία και κάτι πρέπει να γίνει για να ανατρέψουμε αυτή την πορεία. Θέλω να επισημάνω ότι οι έλεγχοι για τους χρόνους οδήγησης και αναπαυσής, δηλαδή οι έλεγχοι των ταχογράφων, τυπικά λειτουργούν βλέπουμε ότι ελέγχονται όλο και περισσότερες εταιρείε, όλο και περισσότερα οχήματα. Αυτό δείχνει ότι ε, οι κόποι της Κομισιόν αποδίδουν καρπούς βεβαίως. Υπάρχουν και τρεις απάτες. Υπάρχουν και απάτες, υπάρχουν και συμπεριφορές, αλλά πρέπει να κινηθούμε σε μια πραγματική κατάσταση και είναι η ιδανική κατάσταση. Αλλά αν δούμε αυτά τα δεδομένα, χρόνια οδήγηση και χρόνια ανάπαυσης, υπάρχει έλεγχος και αριθμητικά ε, βλέπουμε ότι ο έλεγχος γίνεται ε, σε μεγάλο βαθμό, αλλά πρέπει να γίνει έλεγχος και σε άλλες συμπεριφορές, όπως είναι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Δεν τα σε άκουσα ότι είναι στα γαλλικά αυτοί οι εργαζόμενοι. Οι αποσπασμένοι λοιπόν εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται για εβδομάδες και μήνες σε άλλες χώρες, χωρίς να έχουν τα δικαιώματα ε, εργασίας που έχουν οι εργαζόμενοι της χώρας στην οποία απασχολούνται. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί λείπει ο έλεγχος και η εφαρμογή της νομοθεσίας. Δηλαδή το, το νομικό πλαίσιο υπάρχει με την εισαγωγή του ψηφιακού ταχογράφου που μας επέτρεψε να έχουμε πολύ ψηλότερο επίπεδο ε, ελέγχου και τον αριθμό των ελεγχόμενων ημερών εργασίας. Το πλαίσιο λοιπόν υπάρχει. Τώρα πρέπει λοιπόν, να διαβάσω όλα σας τα σχόλια, ερωτήσεις. αλλά ταυτόχρονα με την αύξηση των ελεγχόμενων ημερών βλέπουμε ότι αυξάνεται ο αριθμό των εταιριών που τους επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις. Αυτή λοιπόν η ιδέα ε, ενός μητρώου, ενός αρχείου που να καταγράφει τις εταιρείε ε, στους να βάλουν κυρώσει, είναι κάτι καλό και θα μας επιτρέψει να έχουμε μια βελτίωση της συμπεριφοράς των εταιριών με το πέρας των ε, ετών βεβαίως. Πάντως, αυτή η ανισορροπία και το χάσμα ανάμεσα στις χώρες των 15 και τις χώρες των 12 βασίζεται και οφείλεται σε άλλα προβλήματα και σε άλλα ελλείμματα. Και στις μεταφορές, δηλαδή στις μεταφορές μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα. Αλλά όταν τα πίδα φορολόγησης και τα εισοδήματα διαφέρουν τόσο σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη, τελικά βλέπουμε ότι τα αίτια είναι διαφορετικά σε σχέση με το πρακτικό πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουμε. Σε ό,τι αφορά τις οδικές ενδομεταφορές, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν προτείνω μια διεύρυνση ε, του καμποτάζ. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, το φαινόμενο, να οξυνθεί περιττέρω σε σχέση με την καταγραφή που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σε 10 χρόνια έχουμε μια πολύ χειρότερη εικόνα. Αντί δηλαδή να επιβάλλουμε καλύτερε ρυθμίσει για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, μπορεί να έχουμε μια επιδείνωση ακόμα τη κατάσταση. Okay, can thank you both. Uh, Καλώς σας ευχαριστώ και τους δύο. Σας παρακαλώ να περάσετε στην αίθουσα για να ακούσουμε τους άλλους τέσσερις ομιλητές. Αν νομίζετε ότι εσείς είχατε λίγο χρόνο, αναλογιστείτε ότι αυτοί θα έχουν από πέντε λεπτά ο καθένας. Πιλάρπ, Παλέρο, Νίλσεν Στόξ, Ο κύριος Πιλάμς, ο πρώτος ομιλητής. Okay. Now, gentlemen, five minutes, please. I know... Αγαπητοί κύριοι, πέντε λεπτά ο καθένας, όχι περισσότερο. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλος πειρασμός να ξεπεράσει ο καθένας την ομιλία του το χρόνο τη ομιλία. του, αλλά αυτό βάζει και εμένα στον πειρασμό να πατήσω το κουμπί που σας διακόπτει το μικρόφωνο. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Πίλαρ, έχουμε τον κύριο Πιλέρο από το ETF, ε τον κύριο Νίλσον από την IRU και τον κύριο Στόξ από το Eurocontrol Route που είναι η αρχή ελέγχου. Κύριε Πίλαρπ, θέλετε να ξεκινήσετε εσείς παρακαλώ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ. Ονομάζομαι το Μεπίλαρπ. Είμαι Γενικός Γραμματέας και ε, υπεύθυνο νομικής υπηρεσίας της ε, Σουηδικής ε, Οργάνωσης της, των μεταφορέων και αντίστοιχα εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα ξεκινώντας να δηλώσω και να πω ότι οι μεταφορείς φορτίου δεν ενθαρρύνουν, δεν ευνοούν, ούτε επιτρέπουν συμπεριφορά μη σύνομη, μη σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Τούτου λεχθέντος όμως εντοπίζουμε κάποια προβλήματα ως προς την εικόνα η οποία όπως βλέπουμε παρουσιάζεται με ε, αδρές δεν μας ε, ικανοποιεί και δεν είναι σύμφωνο με την πραγματικότητα. Εμείς ενθαρρύνουμε τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου για τα πλέον εκτίματα και τη δυνατότητα πρόσβαση στην κοινή αγορά. Θέλουμε αυτός ο δημόσιος διάλογος να στηρίζεται σε δεδομένα και πραγματικά περιστατικά και όχι σε φήμες ή συναισθήματα. Ε, ποιον εκπροσωπούμε λοιπόν, μια και έχω λίγο χρόνο, θα σας πω ότι εκπροσωπούμε τους μεταφορείς φορτίου στην Ευρώπη. Πρώτη φορά εδώ, με συγχωρείτε που κάνω λάθος με τις στεφάνιες. Η κατάσταση τώρα. Εκ μέρους των μεταφορέων και πρακτόρων μεταφορών. Και εδώ σημειώνω ότι οι θέσεις μας στερίζονται όχι στην ευρεία έκθεση του φθινοπορού, αλλά στο νοτικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ουσιαστικά τον Ιανουάριο. Η κατάσταση λοιπόν όπως τη βλέπουμε είναι ότι οι πράκτορες μεταφορών, οι μεταφορείς δεν είναι ελεύθεροι να ε, προχωρούν στις μεταφορικές δραστηριότητες. Ε, Υπάρχει περιορισμός σε τρεις δραστηριότητες την εβδομάδα με, με συνέπεια να πρέπει κανείς να οδηγεί το φορτηγό του άδειο ακόμη από τη μία, μέσα σε κάποια διαδρομή ή να, ή να μην μπορεί να φορτώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαφέρουν οι συνθήκες από το ένα κράτος στο μέλλον, στο άλλο. και πολλές φορές χρειάζεται πριν να ξεκινήσουμε τις δραστηριότητε μας να περιμένουμε πολύ καιρό. Οι συνθήκες λειτουργίας λοιπόν διαφέρουν από, τα κράτη, από το ένα κράτος στο άλλο. Σημαντικό πράγμα αυτό και ιδιαίτερα η ενοποίηση φορτίων. Όταν έχουμε τρία-τέσσερα διαφορετικά ε, φορτία με διαφορετικές φορτωτικές από το ίδιο μέρος ε, προελεύσεως στο ίδιο μέρος ε, προορισμού. Δεν μπορούμε να τα συνενώσουμε σε ορισμένε χώρε. Σε κάποιε άλλε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η κατάσταση λοιπόν διαφέρει από κράτο σε κράτο μέλο. Επισημάνθηκε διότι είναι δύσκολο ε, ο έλεγχο εφαρμογή και τη στήριξη των κανόνων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στην αγορά. Προφανώ δεν δεχόμαστε την παραβίαση των κανόνων. Η πρόταση τώρα επί τραπέζης δεν είναι ρηξικέλευθη ε, προσέγγιση η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνεται η ενδομεταφορά ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση, θα έχει δευτερεύουσα λειτουργία σε σχέση με τις διεθνείς μεταφορές και εδώ με τις διαφορετικές στατιστικές που έχουν προβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Eurostat μπορούμε να μιλήσουμε για ένα περίπου 5% αναλογία για τις ενδομεταφορές, ενώ κάποιες άλλες στατιστικές μιλούν για 20%. Οπότε τίθεται το ερώτημα τι μετρούν αυτές τις στατιστικές και πώς γιατί έχω ενδείξεις ότι μερικές φορές χρησιμοποιηθεί το μητρό ε, φορτηγών με ξένη πινακίδα, με ροδοπή πινακίδα και έχουν καταγραφεί όλα αυτά ως ενδομεταφορές, ενώ στην, πραγματικότητα πραγματοποιούσαν διεθνεί μεταφορές. Ε, επίσης, Οι προτάσει ε, με την πρώτη δέσμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας βρίσκουν σύμφωνους για τις 70 μέρες, αλλά όχι τις τρεις μεταφορές, γιατί είναι στην πράξη αδύνατον να επαληθευτεί αυτό και πάση τι σημαίνει μεταφορά. Το τωρινό κανονισμό έχει κάποια προβλήματα, πρέπει να διευκρινιστούν. Επαναλαμβάνω, τι είναι μεταφορά, τι είναι φορτίο, και πώς μπορεί ένα φορτίο ε, να φορτωθεί πάνω στο φορτηγό και να χαρακτηριστεί ως τέτοιο. Υπάρχουν παράνομες πρακτικές τις οποίες θέλουμε και εμείς να καταπολεμήσουμε όπως το ψε, οι ψεύδο ενδομεταφορές, ψεύδο καποτάζ δηλαδή, Αν αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει η ύπαρξη ορισμένων παραβάσεων, δεν πρέπει να παρεμποδίσει την περαιτέρω απελευθέρωση του τομέα. Και τα δύο μπορούν να προχωρήσουν εκ παραλίλου. Ένα ευρωπαϊκό μητρό των, Ευρω... των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, πολύ ευχαρίστω. Δεν δουλεύει το. Τηλεχειριστήριο. Θα προχωρήσω λοιπόν, θα τα καταφέρω, ναι. Έχει λήξει και ο χρόνος. Ε, βλέπουμε λοιπόν από τη δική μας σκοπιά και θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η θεμελιώδης ιδέα βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελευθερία των μεταφορών, της διακίνησης εμπορευμάτων και ε, υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν εμπόδια σε αυτή την Θέλουμε να μπορούμε να αποφεληθούμε αυτή τη αρχή τη ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και εν προκειμένου υπηρεσιών. Τούτου λεχθέντος βεβαίω όλα τα συστήματα θα πρέπει να είναι ε, θεμητά, δεν πρέπει να γίνονται καταχρήσεις της εργασίας των εργαζομένων στο σύστημα αλλά δεν χρειάζεται να αναμένουμε την 100% εναρμόνιση των κανόνων πριν προχωρήσουμε στην απελευθέρωση. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ε, βήμα το βήμα με ένα πρώτο πακέτο μέτρων, με την ε, περίοδο της εβδομάδας των 7 ημερών και μέσα σε, μια, ε, σε ένα διάστημα ενός, δύο, τριών ετών σταδιακά να προχωρήσουμε στην εναρμόνιση. Και έτσι έχω μια ερώτηση προς το Κοινοβούλιο. Γιατί η διεύρυνση φαίνεται να έχει οδηγήσει σε επιδείνωση των συνθήκων, όπως είπαν ορισμένοι. Γιατί κάποιοι λένε δεν μπορούμε να, να ανοίξουμε το σύστημα γιατί θα επιδεινωθεί. Δεν είναι δυνατόν με την ε, διεύνηση του συστήματος να εναρμονηθεί και να λειτουργήσει καλύτερο σύστημα. Εάν είναι έτσι, κάντε το λοιπόν. Ευχαριστώ. Mm. I Ξέρω ότι σε πέντε λεπτά είναι δύσκολο να τα καταφέρετε, το αντιλαμβάνομαι, ναι. Ο κύριος Περίλο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αργαζομένων ε, Μεταφορών. Ρομπέρτο Παρίλο ονομάζομαι και είμαι πρόεδρος των Ευρωπαίων ε, Οδηγών Φορτηγών και εκπροσωπώ όλα τα σχετικά συνδικάτα. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφερθώ σε κάτι που ρώτησα κάποιους ευρωβουλευτές. Κατά πόσο υπάρχουν λύσεις. Ναι, λύσεις υπάρχουν και μπορούμε και να τις θέσουμε σε εφαρμογή υπό τον όρο όμως να ακούσουμε τους επαγγελματίες του κλάδου, δηλαδή τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Θα αρχίσω λοιπόν με την δήλωση των κοινωνικών εταίρων. Είναι σημαντικό να επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή εργαζόμενους και επιχειρήσεις, και έχουμε καταλήξει και σε κοινή θέση και σε κοινή ανάλυση, σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έχουμε και εμείς προτάσεις κοινέ μεταξύ μας. Υπογραμμίζω λοιπόν ότι είμαστε υπέρ μιας αγοράς με θεμητό ανταγωνισμό, χωρίς κοινωνικό ντάμπινγκ. Θέλουμε τα πράγματα να γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά με κανόνες και να τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Σίγουρα θα πήρατε τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων. Μία θέλω να υπογραμμίσω, πολύ σημαντική για μας και που λέει ότι θέλουμε να έχουμε ρυθμισμένη αγορά. Πρέπει να υπάρχει ένας δεσμευτικός χάρτης πορείας, ο οποίος να αναφέρεται στην εναρμόνιση των φορολογικών κανόνων, των κανόνων ασφάλειας, της κοινωνικής ασφάλειας και της εφαρμογής των κανόνων αυτών. Θέλουμε αυτός ο χάρτης πορείας να περιλαμβάνει ένα κατάλογο πρωτοβουλειών, νομοθετικών και μη νομοθετικών, που να επιτρέπουν τη βελτίωση της εναρμόνισης και τη δημιουργία ενός μηχανισμού που να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αντιλαμβάνονται ποια είναι η κατάσταση στην αγορά μεταφορών εμπορευμάτων οδικός και να γνωρίζουν επίσης το βαθμό εναρμόνισης. Όλα αυτά αντιστοιχούν βέβαια σε αυτά που εσείς ευρωβουλευτές έχετε αποφασίσει. Το Νοέμβριο του 2011 εσείς ε, πήρατε μια θέση απέναντι στη Λευκή Λίβρο, ε, και η θέση σας αυτή κάνει ρητά μνήα στη στρέβλωση του κανονισμού και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αναφέρεστε επίσης στην τοποθέτησή σας αυτή στις προτάσεις που θα πρέπει το 2013 να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη, στον κλάδο αυτό. Αναφέρεστε επίσης εκεί σε προτάσεις οι οποίες να μην οδηγούν σε κοινωνικό dumping. Άνοιγμα υπηρεσιών, αλλά όχι κοινωνικό dumping. Αυτά, λοιπόν, έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ω συστάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά ζήτησε από την Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ δεν θα επαναλάβω τα όσα ακούσαμε ήδη, αλλά θα σας δώσω κάποια νούμερα. Σήμερα η μελέτη που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009, η μελέτη που όπως είπε και κάποιος είναι αρκετά ογκώδης, είναι μια μελέτη η οποία περιλαμβάνει τις κοινωνικές συνθήκες και τις δίκες που επικρατούν στον τομέα των δικών μεταφορών. Και τι λέει, κοιτάξτε λίγο το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά χώρα, είναι σαφές. 33.000 ευρώ στις κάτω χώρες, 12.000 στην Πορτογαλία. Και μιλάμε για την Ευρώπη των 15, έτσι. Ρουμανία 2.900. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες μικρές αλλαγές, αλλά αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θέλουμε. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του 2013 να ετοιμάσει μια σοβαρή έκθεση για την ανάλυση της κατάστασης της αγοράς και για την εξέλιξη των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής νομοθεσίας. Πώς αυτή η κοινωνική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη. Για μας δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά εμείς μπορούμε να ελέξουμε την νομοθεσία και ζητάμε να εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει ήδη σήμερα, χωρίς να φτιάχνουμε καινούργια χωρίς λόγο. Θέλουμε η αγορά αυτή να μπορεί να λειτουργεί με συνοχή, με σαφήνεια, σεβόμενη και τηρώντας τις προδιαγραφές για την εργασία. Αυτά δεν είναι σήμερα εφικτά με την ελευθέρωση και δεν καταλαβαίνουμε, εμείς οι κοινωνικοί εταίροι, δεν καταλαβαίνουμε πώς από τη μια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί τον Νοέμβριο μια συγκεκριμένη θέση και από την άλλη οι ευρωβουλευτές έχουν τη θέση που έχουν και το Συμβούλιο επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας λέει ότι η μόνη λύση είναι η ελευθέρωση. Εμείς θέλουμε καλύτερη εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν σήμερα και η Επιτροπή έχει να κάνει μια επιλογή ή που κάνει λευκή βίβλο για φόρες μεταφορές, βιώσιμες μεταφορές ή να μας πει ότι μπορούμε όπως να είναι να μεταφέρουμε στην Ευρώπη και αυτό δεν έχει καμία επίπτωση. Εμείς οι κοινωνικοί εταίροι έχουμε θέση και νομίζω ότι τήρησε και το χρόνο μου. Τέλος, κεφαλαιόδος σημασία είναι να ξέρουμε ότι νομικά μιλώντας οι Κινέζοι και Φιλιππινέζοι οδηγοί φορτηγών μπορούν ελεύθερα να έρθουν και να δουλέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι το οποίο δεν ακούω να σχολιάζεται καθόλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής από τη Διεθνή Ένωση Ειδικών Μεταφορών, ο κ. Μάικλ Νίλσεν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσπαθώ και εγώ να είμαι σύντομο. Ο IRU χωρισμή τα συμφέροντα λεωφορείων ε, πούλμαν ταξί και φορτηγών παγκοσμίω. Το 80% είναι μικρές επιχειρήσεις. Ε, και άρα αυτό πρέπει να λυθεί υπόψη. Σήμερα οι οδικές μεταφορές θεωρούμε ότι σχετικά με αυτό το τομέα έχουμε ανεπαρκή εφαρμογή των κείμενων κανόνων που οδηγούν σε αθέμητο διεθνή ανταγωνισμό στατιστικά στοιχεία που παραπλανούν. Δεν είναι ε, ορθά τα στοιχεία που αναφέρονται και η νομοθεσία, μάλλον οι ε, φορείς, μεταφορείς που ακολουθούν και σέβονται νομοθεσία, αντιμετωπίσουν τον μεγάλο ανταγωνισμό ε, και υπάρχουν πολλά κενά στην νομοθεσία που εκμεταλλεύονται κάποιοι. Έπειτα, η κρατική πολυτροπική σε αυξάνουν την πίεση για τη μείωση των τιμών. Και αυτό το κάνουμε το κυβερνητικό χρήμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα, αποτελεί ζήτημα, διότι υπάρχει και τόσο μεγάλη πίεση για να μειωθούν ε, οι δαπάνες των μεταφορών, οι τιμές των μεταφορών, όπου σε κανένα περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε απόλυτα για ασφάλεια και οικολογική συμπεριφορά, αλλά και για σωστές συνθήκες εργασίας πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον νομικό περιβάλλον με ένα ε, για όλους. Το μέλλον τώρα των ενδομεταφορών θέτουμε ένα αμφιβόλο σημαντικά την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, αναθέρωση μαθησίας. Όλες οι πιθανές α, αλλαγές προτείνει η Κομισιόν ανοίγουν την αγορά σε ένα μεγάλο βαθμό. Α, θεωρούμε ότι η αύξηση της αποτελεσματικότητας που αιτιολογεί η Κομισιόν για αυτή την προσέγγιση δεν ε, θα υπάρξει παρά μόνο περιθωριακά και δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε επιλογή. Κανείς μας πιέζει να κάνουμε κάτι τέτοιο. επίση θεωρούμε ότι το άνοιγμα των αγορών που προτείνει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή θα οδηγήσει σε μια επιδείνωση της όλης κατάστασης ουσιαστικά. Όπως είπε και ο κύριος Παρίλο, και εμείς ως τιμικοί εταίροι προτείνουμε εναλλακτική πολιτική. Πρώτα απ' όλα να διατηρήσουμε το στόχο να μην ανοίξουμε περισσότερο την αγορά, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των κείμενων κανόνων και να ορίσουμε έναν οδικό χάρτη για περισσότερη εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσία. είναι κάτι που ελέγχεται και από την ΕΣΥΑΡ. Για να κλείσω, προσπαθώντας να τηρήσω το χρόνο που μου έχετε δώσει, θέλω να πω ότι είμαστε της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει πραγματικά να κάνει κάτι, και αυτό ελπίζουμε να το υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να δεχθεί την πρόταση των κοινωνικών εταίρων στον τομέα των οδικών μεταφορών κάτι που δεν βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα. Επίση θα πρέπει να βασίσει μια πιθανή τη πρόταση Κομισιόν. Αν τελικά κρίνει αναγκαίο να υποβάλουμε και από αμφιβάλλουμε την αναγκαιότητα για μια νέα πρόταση. Και στην νέα πρόταση, ο, αντί να προτείνει αυτό προτείνει, που για μας είναι ένα πλήρες άνοιγμα των χωρών, καθώς ανοίγει την ε, επιχείρηση σε 7 ημέρες χωρίς καμία εγγύηση, καμία επικλήτα ασφαλείας για τον εργαζόμενο. Η νομοθεσία αναθεωρήθηκε το 2004. 100 από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία ήταν ότι θέλουμε κάποια ποσοτικά μέτρα. Να, γι' αυτό τρεις λειτουργίες αν 7 ημέρες. Και τώρα α, το επιχείρημα και λέτε ότι πρέπει να το άρουμε αυτό γιατί δεν είναι εφαρμοστή νομοθεσία. Ε, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Θα πρέπει να τηρήσουμε την κειμένη νομοθεσία. Δεν υποστηρίζουμε περαιτέρω φιλελευθερωποίηση και άνοιγμα των αγορών. Θεωρούμε ότι ήδη σήμερα υπάρχει στρέβλωση της αγοράς και βλέπουμε ότι οι τιμές συνεχώς συμπιέζονται και θεωρούμε ότι υπάρχει και πιθανότητα ο επαγγελματισμός που διέπει τον κλάδο σήμερα να ε, θυγεί σημαντικά και θα υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση για αύξηση του κέρδους στον τομέα. Άρα δηλαδή θα επιδεινώσουμε την κατάσταση ε, για τους εργαζόμενους χωρίς να παρέχουμε ε, αξιοπρεπής και αυτό δεν αφορά μόνο στους αλλά αφορά την οδική ασφάλεια και την οικολογική συμπεριφορά. Και δυστυχώς δεν είμαστε μόνοι ε, που το πιστεύουμε αυτό. Θεωρούμε ότι όλοι θα πρέπει να είναι υπόλογοι για την εφαρμογή της κύπνης νομοθεσίας και των αναγκών της αγοράς. θεωρούμε ότι μόνο τα μονοπόλια είναι που θα αποφεληθούν αυτές τις αποφάσεις. Ευχαριστώ κύριε Νίλουσεν. Και εν τέλει από την αρχή επιβολής, Φίλιπ Στόξ, Eurocontrol Ρούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Φίλιπ Στόξ και είμαι μέλος του... Χωρίς μικρόφωνο μίλητη. Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεται. Βλέπουμε ότι μπορεί να ληφθεί δράση σε σχέση με όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός είχε γεννήσει πολλές ελπίδες αλλά δεν τηρήθηκε και έτσι πολλές φορές εμφανίστηκε η ανάγκη για ε, έκδοση ή εθνικής είναι ή νέα ερμηνεία της ισχύουσα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Με διαφορετικά επίπεδα λοιπόν εφαρμογή των μεταφορών στα κράτη-μέλη, καταλήγουμε σε μια πολύ σκεχημένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι μεταφορέ στην Ευρώπη αυτήν την εποχή. Στην πραγματικότητα, η ε, τήρηση των όρων, η επιτήρηση μάλλον τη τήρησης των όρων, είναι μια δύσκολη υπόθεση και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιάσουμε στα πράσα, όπω λέμε, τον μεταφορέα. Οι παραβάσεις είναι το να μην τηρηθούν οι κανόνες από τον ε, μεταφορέα περισσότερες από τρεις ε, εργασίες ε, ενθομεταφορών μέσα στην εβδομάδα, να μην έχουν τις σωστές φορτωτικές κτλ. Η άλλη περίπτωση όμως είναι πιο καλά μελετημένη, που ξέρει πολύ καλά τους κανόνες και επιλέγει να κάνει εσωτερικές μεταφορές με σε άλλο κράτος μέλος τακτικά, προσπαθώντας να αποκρύψει αυτές τις δραστηριότητες από τις αρχές ε, επιβολή τη τάξη για πολλές εβδομάδες μερικές φορές χωρίς να επιστρέφουν στην χώρα προέλευση ή χωρίς να ξεκινήσουν διεθνέ ταξίδι, χωρίς αυτό να είναι ε, παράνομο καμποτάζ, αλλά παράνομη λειτουργία, δραστηριότητα. Μια εσωτερική ε, ε, λειτουργία μεταφοράς μέσα σε ένα τρίτο κράτος μέλος συνεπάγεται ή μάλλον προϋποθέτει εγγραφή στο Μετρό του κράτους μέλους. Επομένως υπάρχει διαφορά ως προς το παράνομο καποτάς παράνομη λειτουργία μεταφορών. Στοιχεία για κυρώσει έχουμε πάρει μόνο από 7 κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποια τα οποία επιβάλλουν κυρώσει από 100 μέχρι μερικέ χιλιάδε ευρώ στο κράτος μέλος αναπόκειται να επιβάλλει το, πλήρω το πρόστιμο, αλλά αυτό δεν αρκεί συνήθω για να αποθαρρύνει τον μεταφορέα ώστε να τηρήσει τις προϋποθέσεις. Τότε φτάνει το κράτος μέλος στην κατάσχεση του οχήματο με αποτέλεσμα βράχη πρόθεσμα, αλλά όταν είναι πολύ συμφερούσες οι προτάσεις για τις ε, συμβάσεις των μεταφορών, τότε είναι και μεγάλος ο πειρασμός. Είναι σχετικά όμως μικρό ο αριθμός αυτών των παραβάσεων και έτσι θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι δεν αποτελούν πρόβλημα. Ωστόσο θεωρούμε ότι δεν γίνεται επαρκή καταγραφή και δήλωση αυτών των παραβάσεων. Άρα έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό ε, νομοθέτημα για την εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να εξετάζεται αυτό το σύστημα του καμποτάζ ε, ευρύτερα μέσα στο πλαίσιο ενός θεμητού και σωστού ανταγωνισμού ο ουσιαστικός έλεγχος και του εργαζομένου από τον εργοδότη του και η τήρηση των συνθήκων ε, υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας επιδεινώνεται όταν δεν τηρούνται οι λοιπές ε, προϋποθέσεις για τις ενδομεταφορές. Οι κοινωνικές ε, διατάξεις παραβιάζονται, δεν υπάρχουν περίοδοι ανάπαυσης ή περιορίζονται πολύ σημαντικά. Δεν μπορεί να γνωρίζει το ιστορικό οδήγησης του ενδιαφερομένου και άρα δεν μπορεί ο εργοδότης να γνωρίζει ε, αν είναι ασφαλές να τα αναθέσει ένα επόμενο δρομολόγιο. Ο οδηγός όσο πιο μακριά βρίσκεται από την έδρα του, τόσο πιο μεγάλο κίνδυνο παρουσιάζει για τις οδικές μεταφορές. Μικρές αλλαγές όπως η απάλληψη των τριών, ημερών, των τριών διαδρομών σε καμποτάζ μέσα στο ημέρο και οι ιδιαίτερε συνθήκε για ειδικού, η απάλληψη των ειδικών συνθήκων για ειδικού τομεί μεταφορών αποτελεί κίνδυνο για, την, ε, για υπεραιτέρω επιδείνωση των συνθήκων μεταφορών στο καμποτάζ για τα οχήματα και του οδηγού. Έχει σταθεροποιηθεί λοιπόν σε ένα βαθμό η αγορά, υπάρχει σε ένα βαθμό ε, οργανωμένη και λειτουργούσα αγορά μεταφορών και ίσως μπορεί να ε, προκύψουν δυνατότητες για περαιτέρω διεύνηση αγοράς, αλλά μόνο όταν εφαρμοστούν σωστά οι καρόνες. Ευχαριστούμε πολύ. Κουν, Μπαχ, Λαπάρμα κτλ. Ένα, ένα λεπτό. Ζέλερ, Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ, Μπράιν. Ευχαριστώ πολύ τους κυρίους ε, Πίλμαρ, Περίλου, Νίλσεν Στόξ. Πολύ διαφορετική περιγραφή της εικόνας μας έδωσε ο καθένας ως προς την αγορά της, ε, των μεταφορών που βλέπουμε εμείς στην Ευρώπη. Και ρωτώ, το δυναμικό των μεταφορών έχει μετατοπιστεί, ναι όχι, και σε ποιο βαθμό προς τις, μικρέ, προς τις χώρες και Ανατολικής Ευρώπης. Κάναμε μια διάσκεψη στη Γερμανία πρόσφατα με μια ξεκάθαρη εικόνα. Η Ολλανδία που ήταν μεγάλη χώρα μεταφορική πριν από 10 ακόμα χρόνια σημειώνει μετατόπιση των ε, μεταφορικών δραστηριοτήτων προ χώρε τη Βαλτική ή τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και εκεί εφόσον επιτραπεί το σύστημα των ενδομεταφορών προφανώ και ε, αποκρισταλώνεται αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Δεν τηρούνται οι ώρε οδήγηση, δεν εξασφαλίζονται οι ώρε ανάπαυσης, οι συνθήκε τη αμοιβή, οι κοινωνικέ ε, εργασιακέ σχέσει. Όλα αυτά έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια κατάσταση η οποία προφανώ πρέπει να επιληθεί από το ενδιαφερόμενο κράτο μέλο. και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό το διοτάσεως. Και γι' αυτό σωστά λέγεται ότι στο ε, καμποτάζ, χώρες που έχουν υψηλό επίπεδο κοινωνικών προδιαγραφών κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, να χαθούν μέσα σε αυτό το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ε, δεν υπάρχουν όρια, όλο και περισσότερο ε, διευρύνεται το καμποτάζ με ε, θεμητούς στόχους να μην ε, κυκλοφορούν με άδειο φορτίο τα φορτηγά, ε, να υπάρχει πιο ενιαία ρυθμίση κτλ. Αλλά δεν επιτυγχάνεται αυτό και πραγματικά απορώ. Κύριος Μπαχ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς, για συνθήκε εργασία και σχέση μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη. Έχουμε περιθώριο πιστεύω για αισιοδοξία. Υπάρχουν πολλές, πολλά παραδείγματα όπου η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταιρών έχει οδηγήσει σε καλά νομοθετήματα. Προς τον κύριο Παρίλο, καταρχά. και αναφέρθηκε αρκετές φορές ήδη σήμερα, ε, μίλησε για εργαζομένους από τρίτες χώρες που δεν εργάζονται υπό νόμιμες συνθήκες. Αλλά εσείς είπατε ότι υπάρχουν ε, εργαζομένοι που εργάζονται με νόμιμες συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό, πώς το ορίζετε, με βάση ποιους κανόνες κρίνεται η νομιμότητα. Και επίσης, ε, ο κύριος Νίλσεν μας είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες ως προς τη συγκέντρωση στοιχείων από τις επιχειρήσεις. και ταυτοποίηση σε σχέση με επιπέρους οδηγούς. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτή την απουσία στοιχείων σε... και το βαθμό της λεπτομέρειας. Ευχαριστώ. Ντεμπάκερ. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλους τους ομιλητές. Είναι όλοι εδώ πεπισμένοι για το ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για επιπλέον ελέγχους και να αντιμετωπίσουμε τις προβληματικές εκείνες εταιρείε οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες που ήδη ισχύουν και να, αντιμετωπίσουμε να εντοπίσουμε επίσης τις περιπτώσεις ε, εκμετάλλευσης όπου υπάρχουν. Έχω δύο ερωτήσεις. Γιατί πιστεύω ότι μέρος της σημερινής συζήτησης ε, μένει σε ένα επίπεδο αρκετά όριστο. Πρώτον, κοινωνική εναρμόνιση. Τι εννοείται ακριβώς με αυτό. Τι θα εναρμονίσουμε στο επίπεδο του Βελγίου και του Λουξεμβούργου ή θα εναρμονίσουμε στο επίπεδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Και αυτό είναι εναρμόνιση. Ένα αποδεκτό επίπεδο. Αυτή είναι μια συζήτηση όμως που πρέπει να γίνει. Προς το παρόν να κάνουμε ένα πινκ-πονγκ. Αν εναρμονίσουμε και επιβάλλουμε τους ίδιους μισθούς, αυτούς που έχουμε στις χώρες Μπενελούξ, και τις επιβάλλουμε για τους ε, εργαζόμενους στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, απλώς δεν θα έχουν δουλειά εκεί οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι ακριβώς εννοείται με το κοινωνική εναρμόνιση. Δώστε μας κάποια παραδείγματα παρακαλώ. Δεύτερον, άκουσα τη συζήτηση για τις τιμές στον κλάδο. Φυσικά και υπάρχει τεράστια πίεση. Η οικονομική κρίση εξάλλου δεν βοηθάει για να τιμολογούνται οι υπηρεσίες αυτές ικανοποιητικά. Συγχρόνως όμως υπάρχει και ο προστατευτισμός. Διάβασα στην έκθεση, πέρα από τις διάφορες άθλιες ιστορίες, άκουσα, μάλλον διάβασα, για έναν βου, από τη Βουλγαρία που λέει «Εντάξει, ένα μήνα εγώ, τέσσερις μήνες η σύζυγός μου». Και αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας μόνο από τις χώρες της Ευρώπης των 15 βέβαια έχουμε τα στοιχεία αυτά. Απαντήστε μου όμως παρακαλώ και στην πρώτη ερώτηση για το τι εννοείται με την κοινωνική εναρμόνιση. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις τους. Θέλω να ρωτήσω εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάποιος εδώ που εκπροσωπεί την Επιτροπή. Πότε θα έχει μια νομοθετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροποποίηση του κανονισμού 1071 και 1072 του 2009. Στις μελέτες που παρουσιάστηκαν πριν και από αυτά που είπατε εσείς τώρα για το Ευρωπαϊκό Μητρό των Επιχειρήσεων Μεταφορών, δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των μητρών αυτών. Εγώ ρώτησα την Επιτροπή, τέτοιο μητρό θα έπρεπε να διασυνδέεται το 2012. Μόνο η Βουλγαρία είχε ένα ηλεκτρονικό τέτοιο μητρό και μπορούσε να το διασυνδέσει. Και υπάρχουν και άλλες πέντε χώρες που προσπάθησαν να το κάνουν, αλλά δεν το έχουν κάνει ακόμα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 26 και το τονίζω 26 διαδικασίες επιπαραβάσεις σε βάρος χωρών που δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν τη διάταξη για το μητρό αυτό. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Το μόνο που θέλω να πω τελειώνοντας είναι ότι σε περίπτωση και σε περίοδους ε, κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες φοβούνται ότι υπάρχει ένας φόβος αβάσιμος για τις μεταφορές που έρχονται από την Ευρώπη το 2015 εξαιτίας των φθηνών μισθών που λένε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ενδομεταφορές όμως σταδιακά θα οδηγήσουν σε ομοιομορφία συνθήκων και μισθών. Και αυτό ακριβώς είναι που συζητάμε συζητάμε τελικά τον φόβο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Ο κανονισμός όμως του 1072 επιτρέπει στις χώρες μέλη να απασχολούν οδηγούς από τις Φιλιππίνες, για παράδειγμα. Για λιγότερο από 185 μέρες και μπορούν να χρησιμοποιούν ε, τα φορτικά όχι μόνο για τις εδώ αλλά και για διεθνείς μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, καλά θα κάνουμε να αναλύσουμε γιατί επιτρέπεται αυτό από τον κανονισμό 1072 που ενθαρρύνει τελικά την πρόσληψη οδηγών οι οποίοι δεν εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Δεν ε, εκπληρώσουμε ιδιαίτερα με την ε, πορεία που έχει πάρει αυτή αλλά απογοητεύουμε σε το τέτοιο βαθμό. Θέλω να εκφράσω πρώτα απ' όλα κάποιε απόψει ε, για το τι μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα και δεν μα επιτρέπουν να, να τρέξουμε γρήγορα την πιθανή απελευθέρωση αγορά και Ξέρετε, όταν ε, μειώνεται τη μέση λόγω της κρίσης ε, υπάρχει ε, overcapacity, δηλαδή αυτή είναι η βασική κανόνα της οικονομίας. Αν προσπαθήσουμε να κλείσουμε διδάγματα μακροπρόθεσμα, τότε λέτε να σταματήσουμε την απελευθέρωση, να επιβάλλουμε πιο πολλούς περιορισμούς, οπότε θεωρητικά οι πιο πολλοί περιορισμοί οδηγούν σε πιο άσχημες μορφές διακρίσεων. Αντί να έχεις 15, ξέρω εγώ, 20 αγορές χωριστές, λες, τους δίνεις την ταμπέλα Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά λέτε για κοινωνικό dumping εδώ, σε αυτό τον οίκο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι υπάρχει ο κανόνας να α, έχουμε ένα, αν θέλετε, κοινό ποσό ε, για τη γραμματεία, αλλά μπορούμε και να προσλάβουμε 11 Βουλγάρους ε, ή έναν Δανό. Ε, αν θέλετε, το ποσό είναι το ίδιο. Αυτό τι είναι, είναι dumping που κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι απογοητεύομαι από την πορεία που έχει πάρει η συζήτηση. Όχι συγκεκριμένα γιατί μιλάμε για τους μεταφορείς, αλλά για τη στάση που κρατά το Κοινοβούλιο. Ή πρέπει να δούμε ακροπρόθεσμα το θέμα, να δούμε πώς στηρούνται οι τέσσερις βασικές ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να ξεχάσουμε τελείως για ένα μεγάλο διάστημα αυτό το θέμα. Κύριε Λεφτεμπέργκερ, ευχαριστώ πολύ. Οι δύο συνάδελφοι έθεσαν το ζήτημα της κοινωνικής αναρμονηση ήδη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και λόγω των ε, αντιδράσεων της τάσεων των κρατών μελών ε, ως προς τις κοινωνικές ρυθμίσεις απαραίτητο, αλλά το είδαμε και στην ε, οδηγία για την απόσπαση και σε άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να περιορίσουν το κοινωνικό τάμπινγκ ότι υπήρχαν σημαντικές αντιστάσεις και δεν φέρνουν το αποτέλεσμα. Η έλεγχη από πλευρά των κρατών μελών δεν είναι κατάλληλη για να περιορίσουν το κοινωνικό ντάμπινγκ και θα ήθελα να καλέσω τους ε, εκπροσώπους των ε, επιχειρήσεων τι κάνετε στην πραγματικότητα για να περιορίσετε τις ε, παρεμβάσεις. Έχετε στη τελευταία ανάλυση την υποχρέωση να προστατεύσετε τα ε, νομότυπα εντό εισαγωγικών μέλη σας. Επομένως, τι κάνετε, δεν θέλετε να καταγγείλετε τους ε, παραβάτες. Και μια δεύτερη ε, ερώτηση προς τον κύριο το οποίο το όνομα δεν μπορώ να διαβάσω. Είπατε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κατά λάθο παραβιάζει κανείς την ε, νομοθεσία για το καμπατάζ. Πράγμα το οποίο εμένα μου φαίνεται κάπως παράλογο, απίθανο, θα ήθελα να μου το εξηγήσετε, γιατί νομίζω ότι αν κάποιος ξέρει γραφή και ανάγνωση μπορεί να καταλάβει τι λέει το καμπατάζ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Σενάλοβα, όχι. Να ακούσω τους, δύο ομιλητές, τους τέσσερις ομιλητές από δύο λεπτά τον καθένα για να μην ε, κάνουμε έτσι, λάθος κοινωνικούς χειρισμούς, εμείς, να μην είμαστε εμείς οι κακοί κοινωνικοί εταίροι και παραβιάζουμε τους όρους εργασίας των εργαζομένων. Παρακαλώ πρώτα τον κύριο Πιλάρ και παρακαλώ να, απαντήσετε στις ερωτήσεις που απευθύνθηκα σε εσά. Με τη σειρά που μιλήσετε λοιπόν, Πιλάρ πρώτα. λίγο μετά. αν θεωρείτε, χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος, αν θεωρείτε ότι δεν έχετε κανένα σχόλιο να κάνετε, έχει καλός, κύριος Ετσι ETF. Πολύ σύντομα η περίπτωση των Φιλιππίνων που εργάζονται στην Ευρώπη με, σε κάθε νομιμότητα είναι βασισμένη στον ε, κανονισμό 1072 του 2009 ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα πιστοποίηση από τον ε, εργοδότη προς τον μεταφορέα ονομαστικά και η πιστοποίηση αυτή μπορεί να έχει διάρκεια ζωή 5 ετών. Είτε είναι Κινέζο, είτε είναι Βρεζιλιάνο, είτε είναι Φιλιππίνος, μπορεί να έρθει να δουλέψει στην Ευρώπη χωρί πρόβλημα, όπω θέλει, χωρί κανένα περιορισμό και μετά διερωτώμεθα για την κατάρτιση, για το CAP ε, και όλα αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει πάση να απασχολήσει του νομοθέτε και επίση έγινε λόγο για αναρμόνιση και ρωτάτε τι είδους αναρμόνιση, μα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να ένα παράδειγμα. Έχουμε εργαζόμενου, έχουμε οδηγού από τι χώρε τη Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που μένουν στα υπόλοιπα κράτη για μήνε. Αν δείτε όμω την απόφαση της 15 5η Μαρτίου του 2011 ε, του κ. Σκός, του Ευρωπαϊκού ε, δικαστηρίου με βάση την νομοθεσία του 2008 είναι υποχρεωμένο ο εργαζόμενος να διαμένει στη χώρα στην οποία είναι η έδρα του. Ε, νομίζω αυτό είναι το στοιχειοδέστερο. Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνε που υπάρχουν οι κανόνες αυτοί και εφόσον υπάρχουν και βέβαια συνοδεύονται και από, τους σχετικούς, ε, από τις σχετικές κοινορώσεις πρέπει να είναι αρκετά αυστηρές όμως οι κυρώσεις αυτές γιατί αυτός ο οποίος θα κάνει την παράβαση με 2% ε, ελέγχους, μας λέει ότι έχει μόνο 2% πιθανολόγηση να συλληφθεί και ως του να πληρώσει ε, κάποιο πρόστιμο ή να υποστεί κάποια κύρωση. Άρα λοιπόν με τους κανόνες που ισχύουν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά. Οι οδηγοί από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μας το λένε. Μας λένε αυτό που θέλουμε είναι να δουλεύουμε σε καλές συνθήκες εργασίας. Κάθε 15 μέρες ή κάθε 3 εβδομάδες να γυρνάμε σπίτι μας, να μην περνάμε 6 μήνες ολόκληρου στην Ευρώπη, αδιάκοπα. Και αν δεν ε, γίνεται ε, αν όμως δεν γίνεται δεκτό αυτό ε, που μας ζητούν και ζητούμε να γυρνάμε σπίτι μας κάθε τρεις εβδομάδες και όχι κάθε έξι μήνες να βλέπουμε την οικογένειά μας και τα παιδιά μας, τότε δεν μας δίνουν δουλειά. Κύριος Νίλσον. εγώ τουλάχιστον είχα λεπτό να προετοιμαστώ. Κύριε είπατε πιο πολύ Εμεί δεν θέλουμε πιο πολλού περιορισμού. Εμεί θέλουμε του κανόνε που ισχύουν να εφαρμόζονται. τρει ε, εργασίε, τρει υπηρεσίε ε, σε 7 μέρες αυτό δίνει αποτελεσματικότητα. Ποτέ δεν είπαμε ότι δεν είναι αποτελεσματικέ μεταφορές αν λειτουργεί το καμποτάζ με αυτόν τον τρόπο. Α ισχύσουν λοιπόν οι κανόνε που υπάρχουν. Κύριε Κούν, Είπατε για έλλειψη δεδομένων. Ναι, πράγματι και εμείς συμφωνούμε. Υπάρχει έλλειψη δεδομένων που θα μας επιτρέψουν να λάβουμε σωστές αποφάσεις. Χρειαζόμαστε πιο ισχυρά και αξιόπιστα δεδομένα και θεωρούμε ότι κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή για περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και αν γίνει αυτό όμως, έτσι όπως έχει κατάσταση, το μόνο που θα γίνει είναι να επιδεινωθεί με τις αλλαγές. Ακούστηκε επίση μια άλλη ερώτηση για την πίεση στις τιμές και εναρμόνιση των κοινωνικών συνθήκων. Δίκιο έχετε, είναι δύσκολο αυτό, το ε, λέτε από το κοινοβούλιο. Κάπου πρέπει να συναντηθούμε. Κάποιοι πρέπει να μειώσουν τον πύχη των προσδοκιών τους, κάποιοι θέλουν πρέπει να τον αυξήσουν. Μπορούμε να μειώσουμε τον πύχη μόνο σε επίπεδο μισθών. Όχι, ας δούμε και τα τέλη και τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε κάποιες χώρες που είναι πολύ ψηλότερες από άλλες χώρες. Ε, είναι και αυτή συζήτηση που να γίνει. Τι μπορεί να βοηθήσει το θέμα της συμπίεσης των τιμών, αν υπάρχει κοινή ευθύνη, να είναι όλοι υπόλογοι. Όποιος παίρνει μια απόφαση να, ε, για τη μεταφορά να είναι υπεύθυνο για αυτή την απόφαση. Οπότε με αυτή την ε, κοινή ευθύνη να μπορεί να ε, είναι υπόλογος αυτός που αναλαμβάνει την απόφαση κάθε φορά. Ε, ακούστε μια ερώτηση που δεν απευθύνει και σε μένα, αλλά σας απαντώ. Αυτό σημαίνει ότι κανείς, και όχι μόνο οι μεταφορές, δεν θα αναγκάσουν να παίρνουν αποφάσεις που θα προτιμούσαν να μην πάρουν. Εμείς θέλουμε κανένα να παραβιάσει τους κανόνες. Ε, αλλά αν μια εταιρεία δεν έχει κέρδος, όταν κανείς, μιλάμε για μικρό, μικρές ε, πραγματικά επιχειρήσεις που έχουν ένα-δύο υπαλλήλου, ε, δεν βγάζουν χρήμα, έχουν οικογένεια πίσω, ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες. Εγώ μίλησα για τις μεγάλες πολυεθνικές. Αυτές είναι που επιδεινώνουν την κατάσταση και αυτή είναι η επικινδυνότητα του προβλήματος. Ευχαριστώ κύριε Στόρ και κύριο Σπλερ που θέλετε τελικά τα δύο λεπτά Πρέπει να πει και αυτός κάτι. Κύριε Στόρξ, πραγματικό. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, βασιλογή δεδομένων. Η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα που μπορούμε να πάρουμε από τι οδικέ μεταφορέ είναι κάτι που ήδη προβλέπεται στην νομοθεσία. Δεν υπάρχει πολύ σαφήνεια με το πώ θα γίνει αυτό. Και από την οπτική γωνία των μεταφορέων, αλλά και από στους εφαρμόζουν τον νόμο βλέπουν ότι υπάρχει ε, δυσερμηνία του νόμου. Και τέλος, ζητήστε διευκρινήσεις για ένα σχόλιο που έκανα. Κοιτάξτε, κάποιος μπορεί να κάνει αδικήματα στα πλαίσια του καμποτάζ από μη γνώση ή από κακή ερμηνεία των κανόνων. Αυτό μας το έχουν πει ε, και οι οδηγοί. Είναι πραγματικότητα. Υπάρχει και αυτό. Αυτό που εμένα με κλείσει είναι, όπως μας λένε οι ρομεταφορεί για τον κανονισμό 261 και αυτό που σας λένε για τις ορικέ μεταφορές συμπίπτουν. Ευχαριστώ. Λέω Σπίλετ, μου δώσατε λοιπόν τελικά τα δύο μου λεπτά. Δύο λεπτά έτσι, ναι ωραία, ακριβώς. Εγώ θέλω να πω ότι όσοι προωθούν φορτία δεν θέλουν πλήρη απελευθέρωση χωρίς περιβολή ρυθμίσεων. Θέλουμε να κινηθούμε σταδιακά. Αλλά κάπου να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία απελευθέρωσης βαθμιαία από κοινού σε μια εναρμόνιση. Εναρμόνιση στην εφαρμογή των κείμενων κανόνων. Αυτό λέμε και πιστεύουμε ειλικρινά ότι αν ξεκινήσουμε τώρα θα καταλήξουμε σε ένα έρθμο σύστημα. Κοινή ευθύνη. Συμφωνώ. Ε, ε, μάλλον δεν λέω ότι είμαστε κατά, αλλά να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Φοβούμε ότι μπορεί απλά να α, βρεθούμε την πλάτη στον τοίχο. Και σε καμία περίπτωση εμεί δεν θέλουμε να συμβάλλουμε σε αθέμητες μας πρακτικές. Και ακούστηκε μια άλλη ερώτηση. Οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις, τι κάνουν, πώς ενημερώνουν τους για την οδηγία για του προσπασμένου εργαζόμενου. Σα πω τουλάχιστον στη Σουηδία, εμείς ενημερώνουμε τα μέλη του οργανισμού μας, Λέγοντα τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Έχουμε συνεργασία επίσης και με την αστυνομία και με το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Άλλη ερώτηση. Γιατί οι κάτω χώρε δεν είναι πλέον χώρα μεταφορών και έχει μεταφερθεί αυτό το κέντρο στην Ρωμανία. Αυτό δεν έχει να κάνει αγκαστικά με το καποτάζ. Να σου πω τις μεταφορές συνήθως εκεί που είναι το χαμηλότερο εργατικό α, ε, το χαμηλότερο, μάλλον εισοδήματα, το χαμηλότερο μισθό για του εργαζόμενους στα τερματικά. Στα τερματικά και όχι στου οδηγού. Εκεί θέλουμε το χαμηλότερο εργασιακό κόστος. Αλλά δεν κοινωνική κατάσταση. Ευχαριστώ όλους σας θερμά. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Και για μένα τουλάχιστον να κάνω και εγώ κάποιο συμπέρασμα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω ε, είναι όταν πολλοί μιλούν για κοινωνική εναρμόνιση, για εναρμόνιση των κοινωνικών κανόνων. Η κοινωνική εναρμόνιση συνήθω είναι πρόβλημα όταν πρέπει να πάει προ τα πάνω. Όταν πάει προ τα κάτω, κάνει ένα πρόβλημα αλλά φαίνεται ότι τελικά βυθιζόμαστε όλο και πιο πολύ προ τον πάτο παρά να ανεβαίνουμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Αυτό είναι από τα βασικά ζητήματα. Κατά το τελευταίο μου σχόλιο, Τρει αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση που μάλλον έχουν ξεχάσει πολλά πολλά κράτη-μέλη. ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και προσώπων. Τι έχουμε τελικά, κράτη-μέλη που συνεχώς αντίκειται σε αυτές τις αρχές. Η χώρα μου το κάνει στην ελεύθερη κυκλοφορία των ε, προσώπων Πάντα το έκανε. Αυτό όμως είναι μια θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντοτε να ρίχνω ε, το φταίξιμο στα κρατη Τελικά ε, φτάνει τα κρατη Τι να κάνουμε. Φορείς εφαρμογής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είχαμε κάποιον εκπρόσωπο σήμερα εδώ. Λέτε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και στην εφαρμογή. Μα υπάρχουν φορείς εφαρμογής όπου είναι η πολιτική ρεμπορία που πολλοί απλά κάνουν τον πόντιο πιλάτο. Ο καθένας είναι τα σχήρα του. Σκέφτομαι και πάλι το κανονισμό 261. Παρακαλώ, ε, τουλάχιστον να προσπαθείτε να κάνετε κάτι. Αυτά σας ευχαριστώ όλους και τον κύριο Παστόρη και την κυρία Φριζόνη και στους τέσσερις τελευταίους ομιλητές ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Σίγουρα μας επιτρέπει να σκεφτούμε πολλά. Ξέρετε, εγώ δεν είχα σκεφτεί, δεν είχα καταλάβει ότι τα πράγματα είναι τόσο κακά όσο φαίνονται. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Σε ευχαριστώ όλους για τους συναδέλφους. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρία είναι Δευτέρα 6 Μαΐου στις 3 το απόγευμα. Και όσοι επισκέφτεστε τη βορειοδυτική Αγγλία, την επόμενη εβδομάδα θα σας υποδεχθώ και ευχαριστώ θερμά τους ε, διερμηνείς για τη δουλειά τους.